Good morning, colleagues, and Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, πρώτη μετά τις θερινές διακοπές και τις εκλογές. Ξεκινάμε μια κάποια καθυστέρηση, αλλά ελπίζω στο μέλλον να ξεκινάμε πολύ πιο νωρίς, χωρίς καθυστερήσεις συνεδριάσεις μας, γιατί διαφορετικά δεν θα ε, μένει χρόνος για να μιλήσετε εσείς και να σας ακούσουμε. Ελπίζουμε λοιπόν να περάσατε ένα καλό καλοκαίρι μπορούμε να... και έτσι να μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Φρέσκι, φρέσκι. Μπορεί βέβαια να κάναμε διακοπές, αλλά όπως και εγώ φαντάζομαι και εσείς ε, παρακολουθήσατε τις ειδήσει και είναι πολλοί αυτοί στον κόσμο οι οποίοι δεν πέρασαν καλά το καλοκαίρι αυτό, είτε ήταν η Γάζα, είτε ήταν λόγω του Ιουέμπολα, είτε ήταν στην ε, Συρία και το Ιράκ. Έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα τα συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα στον κόσμο, αλλά πάντως έχουμε ευθύνη σε διαφορούς τομείς και περιοχές και θα μιλήσουμε κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια εκεί όπου μπορούμε να την προσφέρουμε και ε, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρασχεθεί ταχύτερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τη Γάζα. Και αργότερα θα έχουμε και την ε, Επίτροπο, την Ευρωπαϊκή Επίτροπο για τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και κυρίως της παροχής της. Ξεκινάω με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Την έχετε λάβει. Υπάρχουν σχόλια, αντιρρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν. Σημείο 2. Έγκριση πρακτικών 7η και 22η Ιουλίου. Εάν έχετε παρατηρήσει, να ενημερώσετε παρακαλώ τη γραμματεία αυτό το τέλο συνεδριάσεω. Εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσει ή παρατηρήσει, εγκρίνονται τα πρακτικά στο τέλο συνεδριάσεω μα. Σημείο 3. Ε, πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών. Έχετε, πιστεύω, το έγγραφο τη 22 Ιουλίου. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις και πάλι ενημερώνεται τη γραμματεία, ιδάλω συγκρίνονται. Σημείο 4, ανακοινώσει τη Προέδρου. Η κυρία ανακοίνωση και ανακοίνωση που έχω γραμματεια ιδαλω ότι προβλέπεται έκτακτη συνεδρίαση τη προεδρου η κυρια ανακοινωση που εχω ειναι οτι προβλεπεται εκτακτη συνεδριαση τη Επιτροπή μα τη Δευτέρα. Προσέχει Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, 4.30 με 6.30 το απόγευμα, με στόχο να συζητήσουμε με τον Επίτροπο Πίμπαλξ, αρμόδιο θέματα ανάπτυξης, για να συζητήσουμε τον στρατηγικό διάλογο και το μέσο για την υποστήριξη της ανάπτυξης, χρηματοδότηση δηλαδή της συνεργασίας, ε, για την οποία έχουμε εμείς αποκλειστικά την ευθύνη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν συμφωνήσει για τα προγράμματα και την χρηματοδότηση και θέλουμε να φτάνουν τα χρήματα στους αποδέκτες τους όπως έχει οριστεί. Αυτό θα είναι το πρόγραμμά μας για την επόμενη πενταετία και ελπίζω να είσαστε όλη τη Δευτέρα, τα απόγευμα παρόντες, για να ακούσετε τον Επίτροπο Πίλμπαξ. Σημείο 5. Ο κύριος Μακουέντι, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι παρόν. Νομίζω θα μας κάνει μια ανακοίνωση από την Επιτροπή. Έχετε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Θέλω να αναφερθώ εν συντομία σε κάποιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα της τρέχουσας Επιτροπής μέχρι το τέλος του χρόνου, οι οποίες θα σας ενδιαφέρουν. Ε, εγκρίνουμε τρία έγγραφα εργασίας για το προσωπικό, είναι η, ανάπτυξη, η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων που έχουν ζητήσει πολλά κράτη-μέλη για μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική και ανθρωπίνη ανάπτυξη και επίσης θέλουμε να επιδιώξουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για την ε, δαπάνες για την ε, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Επίσης θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάναμε πέρυσι για να ε, περαιτέρω αναπτύξουμε το πλαίσιο για την περαιτέρω παρακολούθηση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χρόνο θα κάνουμε, και κάθε χρόνο θα κάνουμε και μια αναφορά, μια έκθεση για τα θέματα του φύλου. Τέλος θα, ε, ε, θα κυκλοφορήσει μια σημαντική έκθεση για τα θέματα υλοποίησης όχι μόνο ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών μελών για τις δεσμεύσεις τους σε θέματα επιστημικής βοήθειας και τέλος, στο τέλος του χρόνου θα γίνει μια πρωτοβουλία για την παγκόσμια εταιρική σχέση για την υποστήριξη του πλαισίου 2015 του χρόνου και την σχετική ε, πρωτοβουλία που θα γίνει του χρόνου για την χρηματοδότηση, για την ανάπτυξη. Ε, θα έρθει και ο ίδιος ο Επίτροπος την ερχόμενη εβδομάδα, όπως είπατε και εσείς, για να σας ε, μιλήσει περισσότερο για, αυτό το, για αυτή τη σημαντική ανακοίνωση. Αυτά από πλευρά μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μακουέιτ. Τώρα, ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι όλα ξεκάθαρα, σαφή. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε την ε, ανακοίνωσή σας και θα δούμε αν χρειαστεί να γίνει κάτι από πλευράς μας. Τώρα περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σήμερα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ματίας Μπερτσάρδ, ο οποίος ε, είναι ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του UNRWA, για την, ε, ε, τις οργανώσεις αρρωγής. Επίσης θα ακούσουμε τον Jean-Louis de τον ε, στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Η ιδέα εδώ είναι να συζητήσουμε το θέμα της Γάζας και πιο συγκεκριμένα τους τομείς που έχουν σχέση με, τις, με το έργο μας, δηλαδή την ανθρωπιστική βοήθεια. Φυσικά το καλό είναι ότι τώρα ε, υπάρχει η κατάβαση του πυρός, η οποία μια... αλλά το κακό είναι ότι πάνω από 2.000 Παλαιστινοί ε, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 60 Ισραηλινοί συμπεριλαμβανομένων και πολλών στρατιωτών διάβασα ότι από τους 2.000 ε, ε, Παλαιστινίους που έχασαν τη ζωή τους, ε, ο νεότερος ήταν 10 ημερών. Και επίσης συζήτησα με τον κύριο Μπέρτσαρντ και θα θυμόσαστε τους εργαζόμενους της UNRWA που σκοτώθηκαν το καλοκαίρι, κάποιο από το προσωπικό που βρίσκεται εκεί. Πρέπει να μην ξεχνάμε το θάρρος των ανθρώπων αυτών που εργάζονται εκεί, να συνεχίσουν, που συνεχίζουν να εργάζονται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Και κάποιοι από αυτούς τους εργαζόμενους, ε, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένα που έχασε τα παιδιά του στην ε, σύγκρουση αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί και πιστεύω ότι ο κύριος Μπέρτσαρτ θα μεταφέρει στους συναδέλφους του τις ε, σκέψεις μας ε, και την συμπάθειά μας προς τα άτομα αυτά. Τέλος θα ακούσουμε αυτούς και μετά θα ε, μιλήσετε εσείς, θα πάρετε το λόγο. Φυσικά δεν μπορούμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα, αλλά είναι καλό να δούμε τι μπορεί να γίνει και πού θα, πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπέρτσαρτ από την Ουνουρουά, ο οποίος θα μας πει από πλευράς του τι συμβαίνει εκεί, επί τόπου αυτή τη στιγμή και επί τη ευκαιρία. Προφανώς πολλά συνέβησαν τον Αύγουστο και κάποια στιγμή ε, συζητήθηκε να συγκληθεί το Κοινοβούλιο για να συζητήσει του θέματος. Όμως έγιναν επαφές μεταξύ της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και της δικής μας Επιτροπή το καλοκαίρι και ελέγξαμε ότι τίποτα δεν υπήρχε που να εμποδίζει την διεκπαιρέωση της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να χρειάζεται σύγκληση του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό οι συναντήσεις έγιναν τηλεφωνικά και έγινε μια ειδική συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα στην οποία, στην οποία κάποιοι από εσά μπορέσετε να παρευρεθείτε. Λοιπόν, κύριε Μπάτσατ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε με την άδειά σας. Θα σας δείξουμε κάποιες εικόνες για να δείξουμε πώς έχουν τα πράγματα και να διαμορφω... θέσουμε το πλαίσιο της συζήτησης. Δύο λεπτά μόνο. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Ένας από τους φωτογράφους μας έστειλε τις φωτογραφίες για να σας τις δείξουμε για να αποκτήσετε μια εικόνα αυτών που θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ που ε, μας επιτρέψατε να σας δείξουμε. Κύριε Πρόεδρε, ε, επειδή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας ε, ε μετά την ε, εκλογή σας και τη συγκρότησή σας ως Επιτροπή. Θέλω να σας συγχαρώ ε, για την εκλογή σας και ως μέλη της Επιτροπής και ως μέλη του Κοινοβουλίου και να σας πω ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις οργανώσεις αρρωγής προβλέπει στην συνεργασία μαζί σας η οποία θα είναι εξίσου καλή πιστεύουμε όσο και με το προηγούμενο κοινοβούλιο. Θα ήθελα με δύο λόγια να πω τι κάνει η οργάνωσή μας, η UNRWA συνήθως. Ε, βεβαίως υπάρχει τώρα η τρέχουσα κρίση στη Γάζα, η, η κατάσταση όμως αυτή είναι θλιβερή και εξαιρετική. Ε, το πλήρες όνομά μας ε, είναι η ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τις οργανώσεις αρρωγής και τα έργα για τους Παλαιστινίους ε, προσφύγους στην ε, Εγγύης Ανατολή. Και σκοπός μας είναι να προσφέρουμε βοήθεια και προστασία σε ε, Παλαιστίνιους πρόσφυγες που φτάσουν φτάσει πλέον τα 5 εκατομμύρια και ζουν στην Παλαιστίνη, την Ιορδανία και στη Γάζα. Δεν έχουμε εντολή να βρούμε ε, λύση στο πρόβλημα. Ε, η εντολή, το καθήκον που έχουμε είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες. Η λύση επαφίεται σε άλλους οργανισμούς. Όμως είμαστε μοναδικοί υπό την έννοια ότι προσφέρουμε βασικές υπηρεσίες. Παιδεία, βασικές υπηρεσίες υγείας ε, και, και πρόνοιας. Και είναι παρόμοιες με αυτές που συνήθως προσφέρουν οι κυβερνήσεις. Επίσης, Έχουμε 13.000 υπαλλήλους στην Μέση Ανατολή για όπου ζουν, στις περιοχές που ζουν όλοι αυτοί οι Παλαιστινοί πρόσφυγες. Όμως, Εν αντιθέσει με τις κυβερνήσεις, η χρηματοδότησή μας είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου από εθελοντικές προσφορές. Στη Γάζα έχουμε περίπου 500 μέλη προσωπικού από τους Παλαιστινίους και διεθνή, διεθνές προσωπικό. Και αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν τη βοήθεια που σας περιγράφουμε. Είναι γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικά στελέχη και μηχανικοί. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσέφεραν αυτή την ηρωική υποστήριξη στη διάρκεια της κρίσης και κυρία Πρόεδρε σας ευχαριστώ θερμά που τους αναφέρατε και αναφέρετε το γεγονός ότι ανάμεσα στις φοβερές απώλειες της σύγκρουσης αυτής ε, έχουμε και απώλεια 11 μελών του προσωπικού μας τις 15 αυτές ημέρες. Επίσης, θέλω να αναφερθώ στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όχι μόνο ε, δωρητής κρίσιμη συμμαχία. Ε, είναι μαζί με τον ΟΗΕ ε, μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους δωρητές. 50% του ε, μισθού του προσωπικού μας καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις σας. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θέμα αυτό για μας και βεβαίως εσείς πρέπει να ενδιαφέρεστε για το πώς λειτουργούμε. Όταν δείτε τι έχει κάνει το προσωπικό μας θα διαπιστώσετε ότι η επένδυσή σας ήταν πολύ αποτελεσματική. Τώρα, ε, ε να επανέλθω στο θέμα της κρίσης. Ε, μια σύντομη εικόνα της κατάστασης πριν από την κρίση η λωρίδα της Γάζας βρισκόταν ήδη σε φοβερή κατάσταση πριν από την κρίση. Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ήταν ανησυχητική. Ένα παράδειγμα, το 2000, το έτος 2000 είχαμε 80.000 άτομα στη Γάζα οι οποίοι στηρίζονταν στην επιστημιστική βοήθεια που προσφέραμε για την επιβίωσή τους. Τον Ιούνιο ήταν 830.000 οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες που στηρίζονταν στη δική μας βοήθεια και είχαμε και 150.000 που υποστηρίζονταν από άλλο οργανισμό. Έτσι, από τα 1,7 εκατομμύρια, το ένα περίπου εκατομμύριο άτομα εξαρτώνταν αποκλειστικά από τη διεθνή βοήθεια για την επιβίωσή τους. Το 65% του, γενικού, του συνολικού πληθυσμού της Γάζας είναι κάτω από 24 ετών. Η ανεργία ήταν στο 40%, η ανεργία των νέων 65%. Και μπορώ να σας δώσω πολλά άλλα στατιστικά στοιχεία. Όμως, επιπλέον, έχουμε κάνει και μια έρευνα που δείχνει ότι το 90% του νερού στη Γάζα δεν είναι πόσιμο. Πράγμα που κάνει την λωρίδα της Γάζας το 2020, όπως υπολογίζουμε, ένα μέρος που δεν θα μπορεί κανείς να ζήσει εάν δεν ληφθούν δραστικά μέσα, ε, μέτρα για να αποκατασταθεί η κατάσταση. Και όλα αυτά πριν από την κρίση. Στη διάρκεια της κρίσης, για να σας υπενθυμίσω μόνο τα πράγματα, εμείς προσφέραμε καταφύγιο σε 300.000 άτομα σε 85 σχολεία. Αυτός είναι ένας πληθυσμός που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της Βόνης, παραδείγματος χάρη. 300.000 μέσα σε σχολεία. Δεν είναι σχολεία όπως τα φαντάζεστε, όπως τα γνωρίζετε εσείς, με ε, λουτρά και άλλες εγκαταστάσεις που έχουν τα σύγχρονα σχολεία. Είναι σχολεία που έχουν βασικές μόνο εγκαταστάσεις, ας πούμε 10 τουαλέτες περίπου. Και κατά μέσο όρο εκεί σε κάθε σχολείο ήταν 3.500 άτομα. Επιπλέον, βοηθήσαμε 40.000 άτομα στα κρατικά σχολεία. Και επιπλέον, μαζί με το WFP, βοηθήσαμε άλλα 5.000 άτομα που είχαν χάσει τα σπίτια τους και δεν είχαν άλλα μέσα επιβίωσης. Συνολικά λοιπόν στην κορύφωση της κρίσης από το 1,7 εκατομμύρια, το 1,6 εκατομμύριο ήταν απολύτως εξαρτημένο από την βοήθεια του συστήματος Ηνωμένων Εθνών, κυρίως της UNRWA, μαζί φυσικά με την ICRC και άλλους. Αλλά βασικά η δική μας υποδομή ήταν αυτή που έφερε το βάρος. Φυσικά ε, ορίσαμε νοσοκομεία και άλλες ε, εγκαταστάσεις, τους τροφοδοτήσαμε με κάψιμα και κάναμε ό,τι μπορούσαμε όσο ήταν αυτό δυνατόν και εφικτό. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι επανελήφθη κάτι λυπηρό. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επλήγει η Γάζα το 8 και το 9 ε, ε, ε, και το 2012 επλήγει και πάλι. Το γεγονός είναι ότι σε όλες αυτές τις κρίσεις ο πληθυσμός της Γάζας είναι ο μοναδικός πληθυσμός στον κόσμο που δεν του επιτρέπεται να περάσει τα σύνορα, να διαφύγει. Ζητήθηκε από τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους και να αναζητήσουν στέγη κάπου αλλού στη Γάζα. Δεν τους είπαν όμως σε ποιο σημείο στη Γάζα. Θα πρέπει επίσης και πάλι να πω ότι όπως και στις προηγούμενες κρίσεις οι εγκαταστάσεις των ομένων εντρών επνίγησαν πάρα πολλές φορές ότι ήταν γνωστά τα σημεία που βρίσκονται από το Ισραήλ. Οι συντεταγμένες του GPS είναι γνωστές στους Ισραηλίτες στρατιωτικούς και τους δόθηκαν σε πάρα πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μαζικοί βομβαρδισμοί έπληξαν αστικές περιοχές, πνικνά, πικροκατοικημένες. Η, ε, στη Γάζα έγινε αυτό και βεβαίως υπήρξαν πάρα πολλά θύματα. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα λυπηρά αυτά δεδομένα, τα είπατε εσείς εξάλλου κυρία Πρόεδρε, αλλά οι άμαχοι στην ε, Γάζα ήταν εκείνοι που πλήρωσαν το υψηλότερο τίμημα. Πράγματι, 1,7 εκατομμύρια όλη η Λωρίδα έχει πληγεί και έχουν καταστραφεί εκατοντάδες χιλιάδες σπιτικά. Υπολογίζουμε, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι ήδη υπήρξαν πολλοί θάνατοι. Εκτός από αυτό είχαμε 11 περίπου χιλιάδες τραυματίες, σοβαρά τραυματισμένους. Αυτό σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε χιλιάδες τραυματιών από τις προηγούμενες εχθροπραξίες. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για αυτή την κοινωνία. Είναι ένα βάσταχτο φορτίο όλοι αυτοί οι τραυματισμοί. 140.000 άτομα έχασαν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της κρίσης και σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε μια πολύ μεγάλη έλλειψη στέγης, κάτι που ήρθε να προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα από το 2004, όταν το Ισραήλ είχε καταστρέψει πάρα πολλές ε, κατοικίες και καταφύγια. Έχουμε παρουσία σε 31 σχολεία και προσφέρουμε στέγη σε 60.000 εκτοπισμένους. Η όλη υποδομή, το νερό, το ηλεκτρικό, το οδικό δίκτυο, τα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία απαιτούν ε, επισκευή ή έχουν ε, κατεδαφιστεί, έχουν κρεμιστεί σαν αποτέλεσμα των βομβαρδισμών. Την προηγούμενη εβδομάδα θα έπρεπε να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν 240.000 παιδιά. Πραγματικά ελπίζουμε ότι τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν τις 10 επόμενες μέρες να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά. Επιτρέψτε μου επίσης να τονίσω ότι είμαστε η μοναδική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών η οποία έχει μια δορυφορική τηλεόραση η οποία προσφέρει μαθήματα στους, ε, στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Αποκατάσταση. Μόλις ξεκινήσαμε σιγά σιγά να καταβάλουμε προσπάθειες για να κάνουμε ένα ποσοτικό καθορισμό του τι θα κοστίσει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το να κυκλοφορεί κανεί ε, στη Γάζα και από την πλευρά τη Καμά και από την πλευρά του Ισραήλ. Θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να διευκρινιστούν πριν αρχίσουμε την ανοικοδόμηση στις διάφορες περιοχές. Παρόλα αυτά, απλά και μόνο για να σα παραθέσω ορισμένα στοιχεία, γιατί ξέρω ότι σα ενδιαφέρουν από τη στιγμή που είστε Πολιτική ε, ε, Επιτροπή ανάπτυξη, υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση ένα μεγάλο ποσό θα χρειαστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, 280 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια και για τις πρώτες δράσεις, την πρώτη αποκατάσταση δηλαδή των καταφυγίων που επιδέχονται αποκατάστασης και των ε, σχολείων. 111 εγκαταστάσεις της Ούρα έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί. Εδώ μιλάμε για τα πρώτα βήματα της ανοικοδόμησης και εδώ συμπεριλαμβάνουμε βεβαίω και τους μισούς 280 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν σε πρώτη φάση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια προοπτική για το μέλλον. Για την ώρα η πάθη κατάπαυση του πυρός είναι προσωρινή. Θα πρέπει να περάσουμε σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της Γάζας. Και αυτή η λύση μπορεί να είναι μόνο πολιτική. Η διεθνής κοινότητα, και εγώ θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να απευθύνω έκκληση σε εσά να χρησιμοποιήσετε όλε τι δυνατότητε που έχετε ω Επιτροπή για να ενθαρρύνετε την πολιτική ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τους θυμίσετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια επιστροφή, μια επάνωδο στην προτέρα κατάσταση. Αυτό θα ήταν καταστροφικό και θα προκύψει η ίδια κατάσταση μετά από την πάροδο ενός χρόνου. Θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με 1,8 εκατομμύρια κατοίκους στη Γάζα. Τους χρειάζεται μία προοπτική. Υπήρξαν ε, προοπτικές ε, για διακίνηση ε, προσώπων και αγαθών. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Και η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να τύχει της πλήρους στήριξης, να μπορέσει να λάβει και πάλι τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα πρέπει να τους δοθεί η απαιτούμενη στήριξη. Τέλος, δεν θα ήθελα να το ξεχάσουμε αυτό, θα πρέπει να υπάρξει και λογοδοσία για όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας. Υπήρξαν πάρα πολλές παραβιάσεις ε, του διεθνούς δικαίου και εμείς από την πλευρά μας ζητάμε, παζί με όλα τα ενωμένα Έθνη, ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να υπάρξει κάποιος, να αποδοθούν ευθύνε ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, αμάχων και εργαζομένων στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε αυτές τις έρευνες που ξεκίνησαν από τα Ηνωμένα Έθνη σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τι συνέβη σε αυτήν την περιοχή. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Κατάλαβα ότι θα μιλήσετε για θέματα που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό. Και αυτό δεν είναι το βασικό θέμα βεβαίως, αλλά κοιτάζοντας προς το μέλλον θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα κονδύλιο του προπολογισμού που αφορά την Ούνρα και ε, την ε, Παλαιστίνη. Μπορώ να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι οι δεσμεύσει και οι δαπάνες είναι οι ίδιες. Όχι όπως συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου, που ε, είναι ε, ε, μακρόχρονα τα διάφορα προγράμματα και όπου οι εκταμιεύσεις γίνονται σιγά σιγά. Εγώ σας απευθύνω έκκληση από τη στιγμή που ασχολείστε με τον προπολογισμό του 2015 να το έχετε αυτό κατά νου, να γνωρίζετε ότι και η Ούρα και οι αρχές της Παλαιστίνης στη δυτική όχθη Βάζα μπορούμε άμεσα να εκταμιεύσουμε την, γενναιόδορη, το προπολογισμό προπολογισμό σας, τα, τα κονδύλια που θα δώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν συγκινητικές οι εικόνες και η περιγραφή της ε, επίπονης δουλειάς που κάνετε. Τώρα έχουμε τον κύριο Ζων Βεντεπρουγέ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόγραμμα ΕΚΟ, υπεύθυνο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Κύριε Ντεμπριγέ, έχετε το λόγο. Καλώς ήρθατε. Κύριε Ντεμπράουερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη μου παρέμβαση ενώπιον της Επιτροπής σας και ως εκ θα ακολουθήσω και εγώ το καλό παράδειγμα του Ματίας εκφράζοντας τις διαβεβαιώσεις μου για την πλήρη συνεργασία των υπηρεσιών τις οποίες εκπροσωπώ σήμερα εδώ κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Είμαστε στη διάθεσή σας Οπότε θελήσετε να έρθουμε να σας μιλήσουμε όσο συχνά θελήσετε ή κρίνετε απαραίτητο. Και βεβαίως για να σας προσφέρουμε και πέραν των τυπικών αυτών επαφών ή αδίποτε πληροφορία ή στοιχείο που σας ενδιαφέρει για το ζήτημα των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων στις κρίσεις που θα σας απασχολούν. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, το θέρος ήταν πολύ δύσκολο, το θέρος που πέρασε. Θα έχετε την ευκαιρία να το συστήσετε και το απόγευμα σήμερα με την Επίτροπο, κυρία Γεωργιέβα. Οι συνάδελφοι, οι πιο παλιοί, οι μεγάλοι της Επιτροπής στα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας, όσοι αυτοί που έχουν τη μεγάλη πείρα δηλαδή, μου λένε ότι δεν έζησαν ποτέ τέτοια περίοδο που να σημαδεύεται από κρίσεις μεγάλης εμβέλειας όπως αυτή που διανύσαμε και εξακολουθούμε να διανύουμε και τώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει και με συγκλονίζει κυρία Πρόεδρε είναι ότι αυτή η κρίση, όλες οι κρίσεις έχουν προέλευση την ανθρώπινη δράση. Δεν ήταν ούτε σεισμός ούτε τσουνάμι. Ακόμα και η επιδημία του έμπολα που φαντάζομαι θα συστήσετε σήμερα το απόγευμα έχει μεν προέλευση φυσικό φαινόμενο, αλλά οι διαστάσεις τις οποίες έχει προσλάβει οφείλονται και αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην απουσία δράσης, παρέμβασης σε πραγματικό χρόνο, στην πρώτη φάση της ανάπτυξης της κρίσης αυτής, η οποία τώρα προσλαμβάνει διαστάσεις μεγάλης επιδημίας. Και στο πλαίσιο αυτό Πριν από μερικές εβδομάδες αναπτύσσετε μια νέα ανθρωπιστική κατάσταση, αυτή που σας εξέθεσε ο Ματίας, με τόσο εύλογο, με τόσο ε, μεγάλη με τόσο καλές περιγραφές, με τόσο πιστές περιγραφές. Πρέπει λοιπόν να επαναπρογραμματιστούν πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί για την Γάζα το 2014 17 εκατομμύρια περίπου και να επαναπρογραμματιστούν όλα τα προγράμματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες ανθρωπιστικές συνέπειες της κρίσης η οποία διαρκώς επιδεινωνόταν μέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει βέβαια να καταστήσουμε απόλυτα σαφέ, και αυτό θα φανεί άλλωστε μέσα στι επόμενε εβδομάδε, ότι τα χρήματα αυτά διαπανήθηκαν για σκοπού άλλου από αυτού που αρχικά είχαν προβλεφθεί. Δηλαδή, ούτω πιν, σκάψαμε ένα λάκκο, ανοίξαμε μια τρύπα, προκειμένου να καλύψουμε τι κύριε προτεραιότητε και επίγουσε ανάγκε. Υπάρχει μια σειρά πιστώσεων που θα δείτε ότι δεν, έχουν, ότι δεν είχαν ε, δαπανηθεί και αξιοποιήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις μέσα στο καλοκαίρι τον Ιούλιο για 5 εκατομμύρια ευρώ πίστοση. Στην επόμενη εβδομάδα θα εγκριθεί μια πρόσθετη παρέμβαση η οποία παραμένει περιορισμένη ως προς το ύψος της ΜΕΝΑ αλλά πάντως εγγράφεται σε μια γενικότερη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας και θα επανέλθω πολύ σύντομα. Εν ολίγης, μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπιστική παρέμβαση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση της Γάζας, όπως προέκυψε μετά την κρίση και την παρέμβαση του Ισραήλ είναι στα 23 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε δύο τομείς παρέμβασης εστιαστήκαμε, έχοντας υπόψη βεβαίως ότι υπάρχουν άλλες οργανώσεις και φορείς που αναλαμβάνουν δράση σε άλλους τομείς και έτσι εστιαστήκαμε στην υγεία, τις ε, ιατρικές παρεμβάσεις ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου έχουμε ένα ελάχιστο, διατηρούμε το μίνιμουμ των υπηρεσιών υγείας παρά τη μεγάλη καταστροφή των υποδομών στις οποίες αναφέρθηκε και ο Ματίας. Αυτή ήταν η πρώτη ε, παρέμβαση, ο πρώτος τομέας παρέμβασης και ο δεύτερος είναι αυτός που έχει να κάνει με το λεγόμενο wash, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγιεινή, την παροχή πόσιμου νερού και ούτω καθεξής. Εταίροι μας είναι ο, ε, η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, η UNRWA βεβαίω, αλλά και το Παγκόσμιο Επιστηστικό Πρόγραμμα με μεγάλες παρεμβάσεις. Κυρία Πρόεδρε, εάν τυχόν δεν το έχετε ακόμη λάβει, μπορούμε να σας διαθέσουμε την τελευταία έκθεση της ε, ανθρωπιστικής μας παρέμβασης της 26 Αυγούστου που θα σας δώσει πιο λεπτομερή στοιχεία για τον τύπο της υποστήριξης που προσφέρουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά όπως πάντα, κυρία Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι, όπως τον έχουμε να κάνουμε με μια κρίση που αποδίδεται ή εντείνεται από την ανθρώπινη δράση, όπως θα σας εκθέσει φαντάζομαι και η κυρία Γεωργίευα, Βεβαίω η παρέμβαση μπορεί να κριθεί με βάση το ύψο της χρηματοδότησης, αλλά πάνω απ' όλα σε σχέση με τις διευκολύνσεις προς πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια που διαθέτουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς, οι φορείς μας, οι εταίροι μας να έρθουμε απευθεία σε επαφή με τον πληθυσμό που βρίσκεται σε δυσκολία. Και εδώ ακριβώ η κρίση που διανύουμε, που διανύσαμε και ξεκολουθούμε να διανύουμε, σηματοδοτείται από μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση γιατί είτε δεν υπάρχει πρόσβαση, ουδεμία πρόσβαση, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Γιατί μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου μπόρεσαν οι ειδικοί μας να μπουν στην λωρίδα της Γάζας. Ένας από τους ε, κύριους εταίρους, η Oxfam του Ηνωμένου Βασιλείου παραδείγματι, έχει πάνω από 30 αιτήσει θεώρησης διαβατηρίου σε εκκρεμότητα οι οποίε αφορούν το προσωπικό τη που θέλει να μπει στη Λωρίδα. Ένα λοιπόν ναι, αυτό, η δυνατότητα πρόσβαση του προσωπικού ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και η ασφάλεια του προσωπικού αυτού όταν πια μπει στη λωρίδα της Γάζας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά κάθε έναν εργαζόμενο στην ανθρωπιστική βοήθεια, είτε είναι εργαζόμενος των ΗΕ, είτε άλλων διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ήταν εσκεμμένη και προφανώς εσκεμμένη η στόχευση εις βάρος των εργαζομένων αυτών της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της σύραξης η οποία έχει τώρα σταματήσει με μια καταπαυση πυρός που ανακηρύχθηκε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε για ε, προβλήματα που συνεχίζονται βεβαίως για ε, ελεύθερους σκοπευτές ή για βόμβες που εξακολουθούν να εκρήγνεται και οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο και οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο και την ζωή ακόμη των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια ή την αποδοτικότητα της προσπάθειάς τους. Όπως είπα, συνεχίζει η προσπάθεια για την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα προσπαθήσουμε να αποδεσμεύσουμε επιπλέον πιστώσεις. Η ανθρωπιστική βοήθεια, ωστόσο, θα έλεγα θα προτιμούσαμε να μην χρειάζεται να παρασχεθεί. Τώρα που όμως πρέπει να περάσουμε σε μια φάση ανοικοδόμησης, αναδόμησης. Ξέρετε ποια είναι η πολιτική, ο πολιτικός προγραμματισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ καλύτερα από ότι εγώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πεπισμένη ότι η επιστροφή στο status quo ante δεν θα είναι η καλύτερη λύση. Του Ναντίον θα είναι η ιδανική συνταγή για να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέψει στη Λωρίδα της να αναπνεύσει, να ξεφύγει από τον αποκλεισμό, να απαλλαγεί από τον αποκλεισμό και έτσι θα πρέπει να συζητηθεί μια ε, λύση που θα οδηγήσει το αποτέλεσμα αυτό. Επίσης ε, υπάρχει μια πρόθεση για μια διάσκεψη των χορηγών κάπου στις αρχές Οκτωβρίου κατά πάσα πιθανότητα. Ο Σωματείας μπορεί να μας δώσει πιο πολλά στοιχεία στο θέμα αυτό. Είναι προφανές πάντως ότι η ανθρωπιστική βοήθεια έχει ή θα ε, έχει πολύ σύντομα αγγίξει τα όρια της και ως εκεί του θα χρειαστεί ένας προγραμματισμός και επαναπρογραμματισμός των δράσεων και κονδυλίων και πάνω απ' όλα της πολιτικής γειτονίας. Έχουμε λοιπόν μικρή, περιορισμένη ορατότητα για το τι έχει γίνει στο θέμα αυτό και από άλλα κράτη-μέλη στην πολιτική δηλαδή διάσταση γιατί και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη δεν είναι σαφές τι είδους παρέμβαση έχει ε, αναπτύξει ο καθένας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε από σήμερα κιόλας χάρη στην πρόσβαση που μπορούμε πια να έχουμε στην Λόριδα της Γάζας, θέλουμε να δούμε τι έχει προσφέρει ο καθένας για να συντονίσουμε τις δράσεις και αυτά για να σταματήσω εδώ, περιμένοντας τις ερωτήσεις βεβαίως των βουλευτών σας, αλλά και για να μην προκαταλάβω τα όσα θα σας πει η Επίτροπος Γεωργίευα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Όλιβα Σότ από την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ που είναι υπεύθυνη για την ε, μακρόχρονη προσπάθεια ανοικοδόμησης. Δεν θα του δώσω το λόγο τώρα, αλλά αφού έχετε το χρόνο να υποβάλλετε εσείς ερωτήσεις μπορεί να του δώσουμε το λόγο. έχουν ζητήσει το λόγο έξι μέλη. Μπορείτε να μου πείτε ποιοι είναι οι υπόλοιποι που θέλουν να πάρουν το λόγο για να δούμε πόσο χρόνο θα δοθεί στον καθένα. 12 άτομα, έχουμε περίπου μισή ώρα. Σας παρακαλώ, δύο λεπτά αναερώτηση. Ε, δύο λεπτά αναερώτηση, ούτως ώστε να έχουν χρόνο να απαντήσουν οι ομιλητές και κατόπιν να δώσουμε το λόγο στη Γενική Διευθυντεύκο. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι ομιλητές, ο κύριος Στία και ο κύριος Νόιζα. Κύριε Στία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τους κυρίους Μισάρ και τους κυρίους Μπρούερ. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις σας. Θα ήθελα να ε, εκφράσω τη θλίψη μας για την ε, απώλεια ζωής των μελών του προσωπικού του ΟΗΕ. Φυσικά όμως αυτό ισχύει και για όλες τις ζωές που χάθηκαν ε, στη διάρκεια αυτής της στρατιωτικής επέμβασης στη Λόρδα της Γάζας Φυσικά έχετε δίκιο ότι η σημασία, για τη μεγάλη σημασία που πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη και ο μεγάλος αριθμός των τραυματιών, πάνω από 11.000. Με δύο λόγια, φυσικά ε, χαιρόμαστε που επετέφθη εδώ και μια εβδομάδα η κατάπαυση του πυρός και θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή στο μέλλον πώς μπορεί να μονιμοποιηθεί και πώς θα μπορέσει να οδηγήσει σε πολιτική λύση, η οποία φυσικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα της ασφάλειας του Ισραήλ. Είναι ένα θέμα που δεν ξεχνάμε από την άλλη φυσικά πλευρά. Ε, έχουμε και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων να αποκτήσουν δικό τους κράτος και την απαραίτητη ασφάλεια και ευημερία, κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας, όπου όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ε, υπάρχει μόνο η τρέχουσα κρίση. Η Γάζα βρίσκεται υποδιαρκή κρίση νομίζω. Είναι ε, μια ε, ενεργή στρατιωτική σύγκρουση αυτή. Εν συντομία τώρα, θα ήθελα να μου μιλήσετε για τον πληθυσμό για την συνεργασία, με συγχωρείτε, με τους βασικούς παράγοντες στην Αίγυπτο και άλλους. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι προβλέπετε ότι θα συμβεί μετά την κρίση αυτή, ώστε να αποφύγουμε να επανέλθουμε ακριβώς στο status quo ante. Ευχαριστώ. Κύριος Νόιβε και μετά η κυρία Χάιτι Χάουφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τους δύο μιλητές. Νομίζω ότι οφείλουμε το σεβασμό στους ανθρώπους που αγωνίζονται στην περιοχή αυτή, εμείς ως Επιτροπή, για τη δουλειά που κάνουν. Έχουμε τώρα να συζητήσουμε δύο πράγματα. Από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς, μέσα στο καλοκαίρι είδαμε κρίσεις στο Ιράκ, τη Συρία, τη Γάζα, τη Λιβύη ενώ το κοινοβούλιο ήταν σε διακοπές. Νομίζω ότι πια δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί αυτό. Πρέπει να έχουμε μια task force έτοιμη να αναλάβει δράση, οποτεδήποτε χρειάζεται να αναλάβει δράση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Πρόεδρο και στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων να ε, επιδιώξει μια λύση που δεν θα επαναλάβει τέτοιου είδους αδράνεια από πλευράς του Κοινοβουλίου. Επίσης, δεν μπορούμε να αποκόψουμε την ανθρωπιστική βοήθεια από μια πολιτική λύση. Πάντοτε και διαρκώς επιδεινώνεται η κατάσταση στην Γάζα. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε ένα status quo, να παγιωθεί δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνει ή μάλλον δεν παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Γάζα, την Παλαιστίνη, την, ε, το Ισραήλ κτλ. Πρέπει να αναλάβουμε δράση και σε σχέση με την Χαμάς. Το λέω αυτό, δεν είναι διαπραγματεύτη. Ε, η Χαμάς για μας δεν μπορεί να κάθεται στους τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί μας, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Σε αυτή την ε, κατάπαυση πυρός η οποία ακολουθεί τον θάνατο όχι μόνο ε, εργαζομένων της ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΕ αλλά και πολλών άλλων αθώων πιστεύω ότι πρέπει να αναζητηθεί ποιος είναι ο υπεύθυνος για αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Και πάλι σε σχέση με τις εξωτερικές μας σχέσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μείνει αδρανείς, δεν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και ελπίζω η νέα εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική να είναι πολύ πιο δραστηρή. Ευχαριστώ η κυρία Χάουταλα. Κύριε Κούσμαν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για το έργο της UNRWA που εργάζεται υπό δύσκολες συνθήκες ε, εδώ και χρόνια και εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό των προσφύγων που πρέπει να βοηθήσετε. Είναι εντυπωσιακό το έργο σας. Επισκέφθηκα τη Γάζα πριν από ένα χρόνο στις λεγόμενους θερινούς αγώνες που υποστηρίζει επί χρόνια η κυβέρνηση Φιλανδίας και μετά την πιο, τον πρόσφατο αυτό πόλεμο ελάχιστη ελπίδα υπάρχει για τα παιδιά της Γάζας. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να, σταματήσει αυτού του είδου, να σταματήσουν αυτού του είδους οι παραβιάσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις πολιτικές μας διαφωνίες και να δούμε το ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό σκέλος. Αυτό που είδα όταν πήγα στη Γάζα είναι ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής μας βοήθειας, διότι χρημα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη ε, χρηματοδοτούμε σε μεγάλη κλίμακα και σε... Ε, τα χρήματα που δίνουμε καταστρέφονται και χάνονται λόγω της βίας. Και θα ήθελα να ρωτήσω και την άποψή σας επ' αυτό, γιατί και οι φορολογούμενοι δίνουν σημασία στις... στην απώλεια αυτής της προσπάθειας. Δεν προτείνω να σταματήσουμε, αλλά να γνωρίζουμε το κόστος αυτής της ε, συνεχιζόμενης παραβίασης, ε, Κάτι άλλο που θα ήθελα να θέσω είναι ότι μονίμως ζείτε υπό την υποψία ότι στηρίζεται τη Χαμάς και ότι ε, φιλοξενείται δραστηριότητες της Χαμάς στις εγκαταστάσεις και εγώ χρειάστηκε πέρυσι ε, να αντιμετωπίσω μια τέτοια κατάσταση κατά την οποία ο Γενικός Διευθυντής σας έδωσε μια ε, λεπτομερέστατη εξήγηση για το ότι δεν ισχύουν αυτά. Αλλά τι έχετε να μας πείτε περί αυτών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπαϊός Κούσμαν και μετά ο Σαλτ Eh, Ευχαριστώ. Μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση. Δεν θα πρέπει όμως ε, να ξεχνάμε ότι δεν επλήγει από τυφώνα, από τσουνάμι, από κάποια φυσική καταστροφή. Η Γάζα καταστράφηκε, σφαγιάστηκε ο λαός από το Ισραηλινό στρατό και από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Η ερώτησή μου είναι τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στο Ισραήλ να δολοφονεί άμαχους ε, παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να καταστρέφεται μια ολόκληρη περιοχή του κόσμου. Θα πρέπει να πούμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δρά όπως δρά αυτή τη στιγμή παραβιάζοντας τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, βομβαρδίζοντας σχολεία της Ούντρα ή νοσοκομεία. Υπάρχει συνενοχή της διεθνούς κοινότητας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώ για συνενοχή γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ε, διεκόπησαν οι εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Υπάρχει μια συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ παρόλο που υπάρχει το άρθρο 2 που αναφέρεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από τις δύο πλευράς. Δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε άλλες περιπτώσεις ε, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην επιβολή ε, κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για την ανοικοδόμηση της Γάζας, για διοχέτευση κονδυλίων κτλ. Ενδεχομένως θα ήταν καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να μην ακολουθήσει τα λεγόμενα από την ενωμένα Έθνη και για να συνεργαστεί με το Παλαιστινιακό λαό κατά της ε, κατάληψης. Κύριε Δεμπρόγκερ, η, ε, ο στόλος της ελευθερίας ότι σε λίγο θα για την ε, ε, Γάζα. Ο στόλος αυτός αποτέλεσε αντικείμενο επίθεσης. νέα ακτιβιστές δολοφονήθηκαν. Θα ήθελα να μου πείτε τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακολουθήσει τις εντολές του Ισραήλ ή θα ασκήσει πιέσεις έτσι ώστε ο στόλος να μπορέσει να φτάσει μέχρι τη Γάζα. Να μην ξεχνάμε σας παρακαλώ όλοι ότι οι, τα στελέχη που βρίσκονται εδώ ε, δεν είναι υπεύθυνοι για την πολιτική ε, αυτό το μας το είπαν από την αρχή. Αυτές είναι, ερωτήσει αυτές είναι ερωτήσεις προς τους υπουργούς, τους Ισπανούς και τους υπόλοιπους. Ο κύριος Γκάρεντ και ο κύριος Κυρλής. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή και εγώ δεν θέλω να μπω σε πολιτική συζήτηση γιατί όπως είπε ο κύριος ε, Μπουσάρ ότι υπάρχει άλλη πολιτική εντολή. Η πολιτική συζήτηση πρέπει να γίνει αλλού. Θα ήθελα να τιμήσω τη δράση της UNRWA εδώ και χρόνια ε, είναι υποδειγματική και συμφωνώ και εγώ ε, ε, ότι πρέπει και η ΕΚΟ και άλλοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να δεχθούν αυτά τα συγχαρητήρια. Μια γενική παρατήρηση. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Θα έλεγα ναι. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος χορηγός, είναι πάντοτε παρούσα, έχει κάνει υποδειγματική ε, παρουσία. Επιμείναμε στην ουδετερότητά μας, την έχουμε στηρίξει. Ε, έχουμε εξασφαλίσει την αντικειμενικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά ε, πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Εμείς ως Ευρωβουλευτές πρέπει να διαρωτηθούμε. Ο οικονομικός προγραμματισμός της επταετίας προσυδειάζει στις συνθήκες αυτές, είναι κατάλληλος για τις συνθήκες αυτές. Όχι, προφανώς. Ήδη είμαστε στο πρώτο έτος Τη δική μου άποψη, όπως είπε η κυρία Χάουταλα, πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρέφονται αυτά που έχουν δημιουργηθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά πάμε και τα ξαναχτίζουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ντεμπρόιερ ή άλλος εκπρόσωπος από την ε, Γενική Διεθνής Ευκό έχει μιλήσει με εκπροσώπους του Ισραήλ για το θέμα αυτό. Ε, θα δώσω το λόγο στους δύο μιλητές για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και μετά θα ακούσουμε την DG DEFCO. Παρακαλώ, ποιος από τους δύο σας θέλει να ξεκινήσει. Ο κύριος Μπέρτσαρτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήταν όλες οι ερωτήσεις πολύ εύστοχες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και τις ομιλήτρες για την υποστήριξη, τουλάχιστον όσους ε, μας υποστήριξαν και για τις ερωτήσεις τους. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Φυσικά κάποιες χρειάζονται πολύ πιο εκτενή απάντηση και πολύ ευχαρίστω μια και τα γραφεία μας είναι αρκετά κοντά εδώ στα κτίρια σας να σας προσφέρουμε επιπλέον και διεξοδικές πληροφορίες εφόσον δεν σας ε, καλύψει πλήρως η απάντηση που μπορώ να σας δώσω τώρα. Ο κύριος Τυρ με ρώτησε για συνεργασία με άλλους φορείς όπως Αίγυπτο, η UNRWA έχει 12.000 μέλη προσωπικού στη Γάζα που ε, ασχολούνται με το 75%, 1,2 δηλαδή εκατομμύρια πολίτες της Γάζας. Δεν έχουμε πολιτική επαφή. Οι πολιτικές επαφές ανήκουν στον Ρόμπερτ Σάρι, είναι αρμοδιότητα άλλου ε, αξιωματούχου των Εθνών, αλλά βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να διατηρήσει την τεχνική τουλάχιστον επικοινωνία και επαφές και με τα Υπουργεία Εκπαίδευσης παραδείγματι γιατί πρέπει να γίνει η προσαρμογή των προγραμμάτων των σχολείων της έναρξης και του τέλους του σχολικού έτους λοιπά Το θέμα για το νερό ή τον ηλεκτρισμό επίσης για την Αίγυπτο, για το Ισραήλ ε, τα πάντα περνάνε μέσα από το Ισραήλ. Για να, οτιδήποτε εισάγεται στη λωρίδα της Γάζας δηλαδή είναι μέσα από το Ισραήλ. Τα σύνορα με την Αίγυπτο τυπικά είναι κλειστά για ε, πολύ μικρά χρονικά διαστήματα εκτάκτος και ε, για άκρος απαραίτητες και επίκουσες ανθρωπιστικές δράσεις μπορούν να ανοίξουν τα σύνορα, δηλαδή αν πρόκειται να περάσουν πρόσφυγες για πολύ χρονικό διάστημα ή και προσκυνητές, αλλιώς τα σύνορα προς την Αίγυπτο είναι κλειστά, οτιδήποτε χρειάζεται εμείς να φέρουμε στη λωρίδα της Γάζας περνάει μέσα από τα νόμιμα συνοριοφυλάκια υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών αρχών. Και φυσικά όποτε στηθεί πραγματογνωμοσύνη μας εμείς προσφέρουμε ε, συμβουλές ή προτάσεις για τα ευρύτερα θέματα χωρίς να μπλεκόμαστε όπως είπα όμως στην πολιτική αλλά αν χρειαστεί συζητούμε και θέματα ευρύτερα που δεν ανήκουν ε, ακριβώς στην εντολή μας. Όπως είπα υπάρχουν άλλοι φορείς και αξιωματούχοι αρμόδιοι γι' αυτά. Η κυρία Χάουταλα έκανε μια ερώτηση, ιδιαίτερος την ευχαριστώ γιατί μου έθεσε το ερώτημα των υποψιών ότι συνδεόμαστε ή υποστηρίζουμε τη Χαμάς. Και εδώ νομίζω ότι έρχεται και η ερώτηση του κ. Γιάνσεν. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε καθημερινά με τέτοιου είδους υπενιγμούς, επικρίσεις εις της Ούνρα. Και πρέπει να σας πω με πάσα τιμιότητα ότι η Ούνρα είναι οργάνωση η οργάνωση η οποία βρίσκεται υπό την πιο αυστηρή επιτήρηση σε όλε τι οργανώσει των ΗΠΑ. Γιατί και εσεί μα επιτηρείτε και οι οργανώσει των προσφύγων και οι χώρε υποδοχή, το Ισραήλ, τα μέσα μαζική ενημέρωση, όλοι οι πάντε κοιτάνε με πολύ μεγάλη προσοχή το τι κάνουμε. Ε, Εμεί λοιπόν την ανάγκη την ποιήσαμε φιλοτιμία. Είμαστε στο δυνατόν πιο διαφανεί στη δουλειά που κάνουμε. Και εδώ ακριβώ, και αυτό νομίζω σχετίζεται με τι δύο ερωτήσει που αναφέρθηκαν, έρχεται το γεγονός ότι είμαστε η μόνη οργάνωση των ΕΕ, η μόνη διεθνής οργάνωση, η οποία κοινοποιεί τον κατάλογο του προσωπικού της σε όλες τις χώρες υποδοχής και το Ισραήλ και όλους τους χορηγούς, δηλαδή και ε, τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Και τους ζητούμε να μας πούν ότι αν έχουν κάποια ανεπιφύλαξη ή ή οδήποτε υπάλληλο, επιφύλαξη, υποψία, υπόνοια, να μας το πει. Το Ισραήλ ούτε μία φορά δεν μας έβαλε ε, ε, υπόδειξη για κάποιον υπάλληλο. Και όμως εμείς παραμένουμε απολύτως αυστηροί στην απόλυτη ανάγκη για αυστηρή ουδετερότητα των υπαλλήλων μας. Και το ελέγχουμε. Και αν ποτέ διαπιστωθεί ότι κάποιος παρεκκλίνει κατά μία τρίχα έστω από την υποχρέωση για ουδετερότητα, έχουμε μια πάρα πολύ αυστηρή διαδικασία να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτό δεν αποκλεί φυσικά το ενδεχόμενο να ε, παρισχρήσει κάποιο στο προσωπικό μα χωρί να διαγνωστεί εγκαίρω. Ακόμη και η Γερμανική Υπηρεσία Υπηρεσιών είχε τέτοιο πρόβλημα με κατασκόπου BND, όπω ξέρετε, η BND. Αυτό λοιπόν, χωρί να το αποκλείουμε, όπω είπα, το αντιμετωπίζουμε με την πιο αυστηρή δυνατή ε, ε, μεταχείριση και με μηδενική ανοχή. Για δε το θέμα της ε, βολής ρουκετών από τα σχολεία της Σούνρα, ακόμη και η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών έχει απορρίψει τέτοιου είδους υπενιγμούς και κατηγορίες. Έχουμε 280 κτίρια, λοιπόν, θα σας πω, 280 σχολεία. Σε περίοδο κρίσεως, πολέμου, βομβαρδισμών, τα σχολεία αυτά, σε περίοδο θερινή, όπως συμβαίνει τώρα, ξέρετε ότι δεν είναι ε, σε χρήση. Είναι κλειστά, άδεια, κλειδωμένα και άοπλοι φύλακες τα φυλάσσουν. Σε μια περίοδο όμως βομβαρδισμού λέμε στο προσωπικό μας να γυρίσει στα σπίτια του, να φροντίσει τις οικογένειές του. Δεν ζητάμε σε κανένα φύλακα να μείνει σε ένα σχολείο άδειο και κλειδωμένο για να το φυλάει. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, όντως υπήρξε ε, παραβίαση της πύλης ενός σχολείου και μπήκαν ένοπλες δυνάμεις μέσα στο χώρο, στο χώρο του. Όταν όμως μειώθηκε η ένταση των μοβαρτισμών, εμείς επιστρέψαμε, ελέγξαμε την κατάσταση, είδαμε ότι υπήρξε παραβίαση του χώρου του σχολείου και αντιμετωπίσαμε ταχύτατα το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει μια task force, μια ομάδα κρούσεως μονίμως εγκατεστημένη στην Γάζα, λέγεται υπηρεσία λειτουργικής υποστήριξης και καθημερινά πρωί βράδυ ελέγχει το παραμικρό, οποιαδήποτε παραβίαση, ακόμη και γραφίτι στους στίχους των σχολείων μας θα ελεγχθούν για να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μπορεί να συμβεί και δυστυχώς και το Ισραήλ είναι αναμεμειγμένος αυτό, γιατί έχει παραβιάσει την ε, αρχή του απαραβίαστου των ΗΕ. Εθνών. Εμείς δεν έχουμε ένοπλους φύλακες για να υπερασπίσουμε τις, ε, τις ομάδες των υπαλλήλων μας, αλλά έχουμε την δημόσια κατακραυγή, την καταδίκη της παραβίασης των κτηρίων και των σχολείων μας ως μέσο άμυνας. Αλλά επαναλαμβάνω, σε καμία απολύτως καμία περίπτωση, δεν υπήρξε επεισόδιο όπου εμείς να έχουμε έλεγχο σχολείου ή κτηρίου και από αυτό το σχολείο ή κτήριο να έφυγαν ε, πύραυλοι ρουκέτες. Αυτό λοιπόν για να δώσετε τις, για να σας δώσω την απάντηση σε ερωτήσεις σας. Αν τυχόν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, θα σας δώσω και πιο πολλά ε, στοιχεία και τεκμηρίωση. Επίσης, ο κύριος Λίτς νομίζω έχει κάνει μια ερώτηση. για τον ε, τρόπο με τον οποίο συμπλέγονται οι στατιστικές για το τι έχει καταστραφεί από τον εξοπλισμό. Οι στατιστικές, όπως σας είπα και εξ αρχής, είναι μάλλον ε, σε αδρές γραμμές υπολογισμοί αυτή τη στιγμή ακόμη. Έχουμε 30% περίπου υπολογίσει ότι η αστική στέγη, η στέγη των αμάχων καλύτερα, των πολιτών, 30% λοιπόν της στέγης των πολιτών έχει καταστραφεί ολοσχερό ημερικός σε κάποιο χρονικό σημείο στη λωρίδα της Γάζας. Το ότι ε, πηγαίνει κάποιος εμπειρογνώμονας να ελέγξει το συγκεκριμένο σπίτι για να πει μπορεί να επισκευαστεί ή χρειάζεται πλήρη κατεδάφιση και ε, ανοικοδόμηση, ακόμα δεν έχουμε φτάσει να το κάνουμε διότι δεν υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας. Άρα έχουμε μία ε, έναν ανδρό υπολογισμό μόνο, υπολογισμό μόνο για το τι περίπου υπολογίζουμε ως ζημιές. Είπα, 30% των οικειών των πολιτών ε, έχουν καταστραφεί. Ξέρετε επίσης ότι υπάρχει σοβαρότατη ε, καταστροφή του, του δικτύου ηλεκτροδότησης των νοσοκομιακών εγκαταστάσεων. Μεγάλο ποσοστό των εγκαταστάσεων της Ούνρα πάνω από όλα τα σχολεία και θα χρειαστούν πάνω από 2 εκατομμύρια για να αποκατασταθούν αμέσως για να μπορέσουν να καταστούν λειτουργικά. Και ως εκ τούτου αυτές είναι εκτιμήσεις τις οποίες μπορώ να σας προσφέρω τώρα Έχουμε την επόμενη εβδομάδα μια διάσκεψη του Αραβικού Συνδέσμου, ο οποίος, η οποία διάσκεψη θα εξετάσει μια πρώτη αξιολόγηση των ζημιών και πιστεύω την επόμενη εβδομάδα ήδη θα είναι διαθέσιμα πιο, πολύ, πιο πολλά και πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Σας παρακαλώ λοιπόν να δείξετε λίγη υπομονή, γιατί δεν μπορώ να δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Για τις έρευνες. Έρευνες έχουν ζητηθεί. Τα Ηνωμένα Έθνη, ε, τον ε, είπα το πρόσωπο του Συμβούλιο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων στη Γενέβη έχουν ζητήσει να διερευνηθεί η κατάσταση. Αυτό μπορούν να κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη, πιστεύω, είναι πάνω από όλα. Αυτό μπορεί να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση, είναι να υποστηρίξει την πρόταση μια τέτοια έρευνα. Έρευνα η οποία δεν προδικάζει αποτέλεσμα ή πόρισμα. Πάνω απ' όλα πρέπει να διερευνηθούν τα πραγματικά περιστατικά. Αυτή είναι η βάση και αυτό λέμε σε όλους όσοι ζητούν να διερευνηθεί η απώλεια ανθρώπινων ζώων και σε όσους έχουν χάσει τους οικείους τους πάνω από όλα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία και μετά να ζητήσουμε την απόδοση ευθυνών. Άρα χρειάζεται πρόσβαση στην τηλεόρυδα της Γάζας, πρόσβαση σε κάθε φορέα παρόντα εκεί και σε έγγραφα. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να υποστηρίζουμε και στην υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Κοινοβουλίου γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ, όσοι συνομιλείτε ιδιαίτερος, να βγείτε από την αίθουσα για τις ιδιαίτερες συνομιλίες σας, για να μην παρενοχλείτε εδώ την συνεδρίασή μας και να ακούσουμε τις απαντήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ και συνεχίζει ο κύριος Μπέρτσερτ για το Ισραήλ. Βεβαίω και θα πρέπει να γίνει μια διερεύνηση του τι έχει ακριβώ συμβεί. Είναι δύναμη κατοχή τουλάχιστον δυνάμει των δηλώσεων των Ηνωμένων Εθνών η UNRWA είναι μέλος των Εθνών. Ο δικός μας ορισμός λέει ότι το Ισραήλ παραμένει δύναμη κατοχής γιατί ελέγχει τη λόρδα της Γάζας, έστω και αν δεν έχει στρατιώτη σε κάθε τετραγωνικό της μέτρο, ελέγχει τον ενέριο χώρο, την, ε, τη χερσαία πρόσβαση αλλά και τη θαλάσσια πρόσβαση, τον ηλεκτρισμό και το νερό, την ηλεκτροδότηση και την ίδρυυση. Άρα υπάρχει ζήτημα ευθύνης. Εδώ και για μας ορόσημο είναι η τέταρτη σύμβαση διάσκεψη της Γενέβης. Στο θέμα αυτό πρέπει με βάση αυτά να γίνει η συζήτηση χωρίς να καταλήγω σε συμπεράσματα. Όταν όμως εγκαταστάσεις των ΗΕ βάλλονται από πειρά που, έχουν, που προέρχονται από την Ισραηλινή πλευρά, ήδη είναι κάπως σαφής η εικόνα. Ο βαθμός της καταστροφής νομίζω το απάντησα αραβικές χώρες. Μας έχουν υποστηρίξει γενναιόδωρα στο ανθρωπιστικό πεδίο. Πρέπει να το πω αυτό, πέραν της γενναιόδωρης υποστηρίξης που έχουμε λάβει από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δικές σας πατρίδες, έχουμε λάβει ταχύτατη και γενναιόδωρη υποστήριξη και από το Κατάρ και από το Ντουμπάι και από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, παραπονιόμαστε. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό υποστήριξης από τα Ισλαμικά κράτη. Ε, σχολικά βιβλία με ε, κατάχρηση στα κείμενά τους. Δεν μπορώ σε αυτό εδώ να δώσω πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν πρέπει να το δικό μας, ε, το δικό μας έλεγχο αλλά πρέπει να σας πω ότι ακριβώς αυτά είναι τα σχολικά βιβλία της Παλαιστινιακής Αρχής τα οποία έχουμε ε, διεξοδικά μελετήσει, ελέγξει, επιτηρήσει. Δεν νομίζω να υπάρχει σχολικό βιβλίο στον κόσμο που να έχουν μελετήσει πιο πολύ ειδικοί. Πέρσι ακόμα νομίζω έγινε μια έρευνα με κάλυψη οικονομική του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Από μια επιτροπή διαφόρων ειδικών, καθηγητών κτλ. που μελέτησαν τα σχολικά βιβλία, τα εγχειρίδια που απευθύνονται στους νεαρούς Παλαιστινίους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ναι, μπορεί να μην είναι τέλεια γιατί ακόμη αναμεταδίδουν και αναπαράγουν κάποια στερεότυπα, αλλά αντισημιτισμό δεν εμπεριέχουν και αυτό είναι σαφές. Πάλι σχολικά εγχειρίδια του Ισραήλ από την άλλη πλευρά αξιολογήθηκαν και εκρίθη ότι χωρίς να είναι τέλεια πάλι να παράγουν μεν στερεότυπα χωρίς όμως να εμπνέουν μίσος κατά των Παλαιστινίων ή των Αράβων. Άρα λοιπόν είπαμε ότι έχουμε να κάνουμε με σχολικά εγχειρίδια που παράγονται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τον τομέα Γάμα ε, για τα παιδιά των Παλαιστινίων που ζουν εκεί. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση του Ισραήλ ανησυχεί τόσο πολύ αυτά τα σχολικά εγχειρίδια, τα παλαιστινιακά, τότε για την επιτρέψη στα αραβόπουλα ε, που βρίσκονται στην επικράτειά της να ε, διδάσκονται. Άρα προφανώς δεν είναι τόσο κακά αυτά τα εγχειρίδια. Γι' αυτό θα σας καλούσα να ακούγεται με πιο μεγάλη επιφυλακτικότητα τις ε, τους μύθους που διαδίδονται για τα σχολικά εγχειρίδια. Ναι, ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία. Η κυρία Μακέιβαν, ναι, έχουμε και την Επίτροπο, ξέρετε, να μας ε, δώσει τις τα υπόλοιπα στοιχεία. Παρακαλώ, κύριος Ντεπχόουερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ζητήσω από το συνάδελφό μου της Γενικής Διάστησης να συμπληρώσει τρία σημεία. Καταρχάς ο προϋπολογισμός. Έχουμε ένα εργαλείο που ονομάζεται απόθεμα έκτακτης ανάγκης ε, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για απρόβλεπτες ανάγκες, για έκτακτες ανάγκες. Εδώ τίθεται όμως το πρόβλημα που ανέφερε ο κύριος Γκέρες στην παρέμβασή του, δηλαδή δημιουργείται μία ε, έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των πιστώσεων δεσμεύσεων και των πιστώσεων πληρωμών, δηλαδή των ποσών που έχουν εκταμιευτεί συχνά η προσφυγή σε, αυτή την, σε αυτό το απόθεμα γίνεται όταν πρέπει, αλλά αναλαμβάνουμε έναν κίνδυνο σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό που μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και σίγουρα η κυρία Γκεργίβα θα θελήσει να το συζητήσει το θέμα μαζί σας. Μπροστά λοιπόν στην σοβαρότητα της κατάστασης το όλο χαρτοφυλάκιο που προβλέπεται στον προπολογισμό ή ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ανθρωπιστικέ κρίσει, ανθρωπιστικέ παρεμβάσει, φαίνεται όλο και περισσότερο ανεπαρκή. Γι' αυτό είναι δραματικό. Πάρα πολύ αναφέρθηκα στην κρίση που καλούμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα δίχως να θέλω να προδικάσω τον διάλογο που θα έχετε με την κυρία Γεωργίευα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο θέματα που από τη μία πλευρά οι ανθρωπιστικές επιτόσεις κρίσης στο Ιράκ που δεν έχουν ακόμα προσμετρηθεί και από την άλλη πλευρά η ανάληψη της σε επίπεδο ε, παγκόσμιο της επιδημίας του ιού έμπολα. Πραγματικά οι πιστώσει που έχουμε είναι στη διάθεσή, στη διάθεσή μας είναι πάρα πολύ περιορισμένες μέχρι το τέλος του χρόνου. Εμείς ε, δεν χρηματοδοτούμε τις κυβερνήσεις. Ε. Συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικού εταίρους και με υπηρεσίες των Ηνωμένων και έχουμε μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου ιδιαίτερα σοβαρούς ε, για να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι μας δεσμεύουν και χρησιμοποιούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως ανθρωπιστική βοήθεια. Τελευταίο σημείο, οι κατεδαφίσεις το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Το πρόβλημα αυτό τίθεται ιδιαίτερα στην περιοχή Γάμα. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα διάλογο με τις αρχές του Ισραήλ. Ματέως, επανερχόμεθα στο θέμα τώρα, η κυρία Όταλα το είπε, ότι αποκλείεται να διακοπεί οποιαδήποτε παρέμβαση γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα ανθρωπιστικό θέμα και θα πρέπει να είναι εκεί. Δεν κοφεύουμε σε ό,τι αφορά το θέμα των κατεδαφίσεων. Πριν από το καλοκαίρι, πριν το ξέσπασμα της κρίσης υπήρξε ένας διάλογος με τις χώρες μέλη σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα εν ώψη της προετοιμασίας νέων μέτρων που θα ληφθούν ως προς το Ισραήλ η νομική οδός είναι και δύσκολη και παρατεταμένη. Θα πρέπει να προβλέψουμε μια πολιτική οδό και στην πολιτική αυτή οδό χρειαζόμαστε όλη την στήριξη όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά όλων των χωρών μελών. Σταματάω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται η Γενική Διευθυντεύκο να πάρει το λόγο, έχουν καλυφθεί όλα τα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τους δύο σας, ευχαριστήσω τους ομιλητές που ήρθαν, που μας αφιέρωσαν το χρόνο, του, τους και που έκαναν μια τόσο ενδιαφέρουσα ανασκόπηση. Υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Θα έρθει και η Επίτροπος. Υπάρχουν και πολιτικά θέματα που θα πρέπει να επιλύσουμε όσο πολιτική και θα πρέπει να αναμένουμε από τους ε, τεχνοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαμε να επιλύσουμε εδώ και είναι ευθύνη μας να τα επιλύσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των διακοπών, είπαμε ότι υπήρξαν διακοπές ε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όλα έγιναν ε, όπως έπρεπε. Βεβαίως ε, δεν θα είχαν επιληθεί τα προβλήματα του προπολογισμού αν είχε συναντηθεί αυτή η Επιτροπή. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια περαιτέρω συζήτηση σχετικά με το τι συμβαίνει σε περιόδους κρίσης. Μια καλή είδηση. Είδα ότι στην Ουκρανία έχει ε, διακηρυχθεί η κατάπαυση του πυρός έχει κηρυχτεί, με συγχωρείτε, κατάσταση του πυρόσα. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία να συνεργαστούμε και πάλι μαζί σας στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Αν κάποιος θέλει να φύγει από την αίθουσα, μπορεί να το κάνει ησύχω. Μπορούμε να περάσουμε στο θέμα 7. Ερωτήσεις. Ώρα των ερωτήσεων. Έχουμε το θέμα, ε, λοιπόν, ε, είμαστε στο 7. Θα ήθελα να πω στα νέα μέλη ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τα μέλη, αν έχουν ερωτήσει για την Επιτροπή, να την υποβάλουν τρει μέρε νωρίτερα και το ερώτημα θα μπορούσε να απαντηθεί εδώ στην Επιτροπή. Βεβαίω, αν υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει, θα πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο τη ημερησία οι άταξη θα συμπεριληφθούν, αλλά είναι μια ευκαιρία για τα μέλη να πούν την άποψή του. Όλοι έχετε αντίγραφο των ερωτήσεων. Δεν θα διαβάσω τι ερωτήσει. Η ερώτηση, πρώτη ερώτηση από τον κύριο Περίνεν και αφορά τη σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Πρώτο το λόγο στον Επίτροπο, μετά στον κύριο και κύριο Δερέινα, αν μπορεί να επιστρέψει, θα κάνει ορισμένα σχόλια. Ο κύριο Σιμονέ έχει το λόγο από την ΤΕΦ. Ευχαριστώ. Και αυτό κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω στη διαθεσή μου, λιγότερο από 3-5 λεπτά. Περίπου τόσο. Θα ξεκινήσω με κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Εν συντομία να σας παρουσιάσω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και κατόπιν τις προπτικές για τη μελλοντική σχέση ε, στο, του αναπτυξιακού διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωμένων Πολιτειών, όπως τον ονομάζουμε για να σας δώσω μια εικόνα της κατάστασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείε είναι κατά πάσα πιθανότητα ο πιο σημαντικός εταίρος μας στη συνεργασία για την ανάπτυξη και ο μόνος που έχουμε αναπτυξιακό διάλογο σε υπουργικό επίπεδο, έναν διάλογο όπου τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν πλήρη ρόλο. Βλέπω ότι κάποια, ε, κάποιοι παρίστανται, κάποιοι συμμετέχονται στο διάλογο. Η λογική της σχέσης μας του διαλόγου και της συνεργασίας ε, ε, ε, μας λέει ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη με τις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν 80% του, της αναπτυξιακής βοήθειας ε, για, ε, που αναφέρεται στον ΤΑΚ. Άρα ε, έχουμε μέσω αυτού του διαλόγου τη δυνατότητα να έχουμε πολύ μεγάλη επίδρα, επιρροή στο χώρο. Ο διάλογος αυτή τη στιγμή γίνεται σε τρία επίπεδα υπουργικό, ανώτερων στελεχών και τεχνικό επίπεδο. Τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Η υπουργική συζήτηση γίνεται μια φορά το χρόνο με τον Επίτροπο, τον Επίτροπο Πίμπαλξ, ο οποίος ε, ε, ε, συνομιλεί με τον ομόλογό του από πλευρά Έχουμε δύο φορές το χρόνο συναντήσει ανώτατων στελεχών και πολλές τεχνικές συζητήσεις για διάφορα ζητήματα. Οπότε, η ερώτησή σας αφορούσε την πρόοδο από τότε που ξεκίνησε ο διάλογος αυτός από το 2009. Πρέπει να σας ε, τιμήσουμε για τον ε, ρόλο που παίξατε ε, στο θέμα της επανέναρξης αυτού του διαλόγου. Από το 2009 λοιπόν, από το Νοέμβριο του 2009 που έγινε η διάσκεψη κορυφής, έχουμε επανενεργοποιήσει τη σχέση μας με τις ΗΠΑ, η οποία όπως βλέπετε αντιστοιχεί με την έναρξη της πρώτης περίοδου Ομπάμα και ε, η πρόταση ήταν να επικεντρωθεί η συνεργασία σε τρεις τομείς, επιστηστική ασφάλεια, ε, ε, κλιματική αλλαγή και MDGs. Ε, αλλά εμείς ε, θεωρούμε ότι ο σημαντικότερος διάλογος είναι αυτός που αφορά την μυστική ασφάλεια και την ε, αντοχή. Όπως γνωρίζετε, οι πολιτικές σχεδιάστηκαν το τέλος του 2012 σε πλήρη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Μπορέσαμε λοιπόν ε, να αλληλοεπηρεάσουμε τις πολιτικές ε, ε, ο ένας του άλλου και αυτό επιτρέπει καλύτερη συνεργασία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγέτης σε αυτή το συντονισμό ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι επικεφαλής, ηγούνται του, ε, της παγκόσμιας πρωτοβουλίας ε, στο κέρας της Αφρικής. Ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε ε, κάποιο άλλο από εμά κάνουμε ε, τίποτα στις περιοχές αυτές, αλλά αποδεχόμαστε ότι ο ένας είναι επικεφαλής στο ένα χώρο και ο άλλος στον άλλον, για να ε, κάνουμε πιο αποτελεσματική την προσπάθειά μας. Μετά θα συζητήσουμε το θέμα των FDGs, MDGs, αλλά έχουμε πολύ καλό ε, επίπεδο διαλόγου με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει μια σύγκληση ε, των προτεραιοτήτων μας για τους αναπτυσιακούς στόχους της χιλιετίας, τους MDGs. Ε, όπως φάνηκε από την διάσκεψη κορυφής, δεν μπορέσαμε να αποδώσουμε πολλά Φυσικά συμφωνούμε με τις ΗΠΑ ε, για τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, μπορέσαμε να συνεργαστούμε στο θέμα της βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής που επηρεάζει τον τομέα αυτό και αυτή τη στιγμή καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες να συντονιστούμε σε αυτά που ε, κάνουν οι πολιτείες ε, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Power Africa και αυτό το που κάνουμε εμείς ε, στα πλαίσια της ενεργειακής εταιρικής σχέσης με την Αφρική. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, έγινε μια διάσκεψη κορυφής ε, φέτος το Μάρτιο. Θα θυμόσαστε, ο πρόεδρος Ομπάμα επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, όπου δόθηκε περαιτέρω πολιτική στήριξη στο διάλογό μας και μας ενεθάρρυνε να επικεντρωθούμε στα θέματα μετά το 2015, στην ανθεκτικότητα, στην ενέργεια, στην Αφρική και την ασφάλεια και ανάπτυξη. Αυτά θα είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε επίπεδο υπουργικών, υπουργών και ανώτατων στελεχών. Υπάρχουν και άλλα θέματα που εμφανίζονται στην ημερήσια διάταξη. Φερρυπίν, η κρίση του έμπολα, ε, αυτό είναι σαφώς ένα θέμα στο οποίο προσπαθούμε να εμπλέξουμε και τις ΗΠΑ για να υπάρξει συνέργεια Τέλος, η μεγάλη ε, πρόκληση θα είναι αυτός ο εκτεταμένος διάλογος πολιτικής να μεταφραστεί σε καλύτερη συνεργασία στην πράξη. Δηλαδή, προσπαθούμε να συντονίσουμε καλύτερα το σχεδιασμό των ε, δράσεών μας σε πιλωτικές χώρες και θα έρθει κάποια στιγμή που θα συζητήσουμε ε, τη φάση της υλοποίησης. Αυτό θα είναι η μεγάλη πρόκλησή μας για το μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την αναφορά αυτή. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα όπως και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό. Υπέβαλα το ερώτημά μου στην αρχή της συνεδρίασης της Συνόδου, γιατί ε, άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το θέμα αυτό δεν έχει ποτέ συζητηθεί στην Επιτροπή. Ο λόγος είναι ότι το 2009 έγιναν οι κοινοβουλευτικές εκλογές. Η πρωτοβουλία μου ξεκίνησε στο τέλος Ιανουαρίου του 2009, έγινε αποδεκτή από το ε, Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης. Τότε ε, Υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο Λουί Μισελ. Υποστήριξε την ιδέα και έγινε αποδεκτή από εμά. Όμως το Κοινοβούλιο ε, ολοκλήρωνε τη θητεία του λόγω των εκλογών και όταν στη Ουάσιγκτον έγινε το Νοέμβριο η συμφωνία για την ε, νέα διάσκεψη κορφής ξεκινούσε το νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Ποτέ λοιπόν δεν υποβλήθηκε μια αναφορά στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Από αμερικανικής πλευράς, ο Μπαράκ Ομπάμα και η Χίλαρη Κλίντον ήταν οι ίδιοι ε, πολύ ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της ιδέας. Άρα έγινε πρόοδος. Ελπίζω ότι μετά το ξεκίνημα αυτό θα έχουμε μια τακτική ε, υποβολή αναφορών προς την Επιτροπή μας για αυτή τη, αυτής της διαδικασίας της συνεργασίας. Είναι κρίσιμη σημασία. Το 80% του λογαριασμού το πληρώνουμε εμείς και η επιρροή μας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη, όχι μόνο στο πεδίο επιτόπου, αλλά και στις διεθνείς ε, διασκέψεις. Ως υπουργό, η εμπειρία μου ήταν ότι το G77 που είναι επικεφαλής η Κίνα πάντοτε διευθύνει, την ορχή, διευθύνει την ορχήστρα και εμείς ε, σε μας ασκούνταν κριτική ενώ είμαστε οι μεγαλύτεροι ε, δωρητές. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στις διεθνείς ε, διασκέψεις. Χαίρομαι που τώρα ε, συζητούνται οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015 σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω απάντηση. Είστε τώρα σε επαφή μεταξύ σας. Ε, και πρέπει να συνεχίσετε την ε, συζήτηση αυτή. Ε, τώρα φτάσαμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τους ομιλητές για την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 θα έχουμε δύο πάνελ, δύο συνεδρίες. Πρώτα οι δύο και μετά οι άλλοι δύο ομιλητές. Πρώτος ομιλητές είναι ο κύριος Μάιρ Χάρτινγκ και ο κύριος Κουμάρ Μπραντέο. Παρακαλώ να ανεβείτε για να αρχίσει η συζήτηση. Και εντωμεταξύ εγώ θα σας παρουσιάσω τη βάση αυτής της συνεδρίασης. Όλοι ξέρετε ότι έχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, τους MDG, οι οποίοι πρέπει να, ολοκληρω... να μέχρι το 2015. Σε πολλούς έχει σημειωθεί πρόοδο, σε άλλους όχι, όμως τα Ηνωμένα Έθνη και η παγκόσμια κοινότητα συζητούν ε, την αντικατάσταση του 2015 και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα το κοινοβούλιο μας πρέπει να εμπλακούν. Το κοινοβούλιο μας πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση. Οι συντονιστέ ε, συμφώνησαν πριν ακριβώ από το καλοκαίρι ότι το κοινοβούλιο μας θα υποβάλει έκθεση δύο πρωτοβουλίε επ' αυτού, η οποία θα ολοκληρωθεί, θα συζητηθεί πριν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, πριν δηλαδή συμφωνήσει τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα την, μετα, την μετατροπή των στόχων για μετά το 2015. Οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν με, από του χρόνου και άρα η ιδέα είναι να ξεκινήσει η συζήτηση ε, να δοθεί στους ε, ευρωβουλευτές η δυνατότητα να ξεκινήσει η συζήτηση. Θα γίνουν και άλλες συζητήσεις, ίσως και μια άλλη ε, ε ακρόαση, έχει ανακοινωθεί και από το ΕΛΚ, ε, οπότε είναι κάτι που θα, κυριαρχήσει στη δουλειά της Επιτροπής μας στο μέλλον. Πολλοί συνάδελφοι είναι νέα μέλη του Κοινοβουλίου και νέα μέλη της Επιτροπής, όπως και εγώ είμαι νέο μέλος της Επιτροπής, δεν γνωρίζουν τι γίνεται ακριβώς στα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα από τη δουλειά μου για την κλιματική αλλαγή, αλλά μην ξεχνάμε, αυτή είναι μια πρώτη συζήτηση εγώ μιλάω για SDGs και MDGs τόση ώρα. Πρέπει να αποφύγουμε ε, την ε, ορολογία αυτή που δεν είναι με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι οι πάντες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τώρα τους δύο μιλητές. Ο πρώτος είναι ο ε, πρέσβης Μέιρ Χάρτινγκ, πρέσβης των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι σημαντικό ε, στοιχείο αυτής της διαπραγμάτευσης, σημαντική προσωπικότητα και κατόπιν θα ακούσαμε από τον πρέσβη Κουμάρ Μπαμπτέο, που είναι ο πρέσβης της Αφρικανικής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ε, κύριε Μάιρ Χάρτινγκ, έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά ο κάθε ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θεωρώ ότι είναι προνόμιο το ότι βρίσκομαι ανάμεσά σας και δεν έχω τη βεβαιότητα ότι είναι τόσο στοιχειώδη τα όσα γνωρίζετε. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά που ξέρουν πολλοί σε αυτήν την αίθουσα. Πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα τη στενή συνεργασία που μπορέσαμε να αναπτύξουμε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα για την ημερησία σας διάταξη. Είχαμε επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της ανάληψης δράσης μου Υπήρξε και αποστολή μία αντιπροσωπεία που δεν ήταν από την Επιτροπή βεβαίως Ανάπτυξης. Είχαμε, συναντηθήκαμε και στο Ρίο και στον, ε, καθώς και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Μπαρόζο στις συζητήσεις ε, και ο επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτσε δίπλα στον πρόεδρο Μπαρόζο. Αυτό δείχνει το πόσο στενή είναι η συνεργασία που έχουμε με το Πρεβικό Κοινοβούλιο. Πριν να μιλήσω για το τι θα συμβεί μετά το 2015. Θα ήθελα να πω δύο λόγια το τι μας οδήγησε στη διάσκεψη αυτή κορυφής. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και Όσο πιο πολύ προχωρήσει η διεθνής κοινότητα, τόσο πιο αξιόπιστοι θα είμαστε για την ανάληψη νέων δεσμεύσεων. Οι επιτροπή συνεργάστηκαν σκληρά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη επιρροή της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι επεξεργαζόμαστε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο μετά το 2015. Δεν σημαίνει αυτό ότι μειώνουμε τις προσπάθειές μας και νομίζω ότι ένα ξεκάθαρο μήνυμα είναι ότι όταν μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα μετά το 2015 η πρώτη πρόκληση είναι να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Ήδη αναφέρθηκα την, στο κομβικό συμβάν της προηγούμενης χρονιάς, το Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης MDG. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το θέμα της εκρίζωσης της φτώχειας και της αηφόρου ανάπτυξης από κοινού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεξεταστούν αυτά τα στοιχεία και θα έλεγα ότι ακόμα και παρακολουθώντας ο κεφαλής της αντιπροσωπείας Εντυπωσιάστηκα με το πώς η ΕΦΚΟ και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος συνεργάστηκαν και μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια κοινή προσέγγιση. Το Ρίο Συνήκωση από την άποψή μας ε, επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση την πρόταση της Επιτροπής εργάστηκαν σκληρά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εμείς στη Νέα Υόρκη ήταν σημαντικό το να υπάρξει μια ηχηρή φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σεπτέμβριο και από τότε συνεχίσαμε τη διαδικασία των ομάδων εργασίας για την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Οι εργασίες αυτών των ομάδων τελείωσαν τον προηγούμενο Ιούλιο. Είπατε κυρία Πρόεδρε ότι ορισμένα από αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρατε, αλλά θα πρέπει να πω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν βίωσα κάτι τόσο πολύπλοκο όσο αυτή η ανοιχτή ομάδα εργασίας. Μια πραγματική πρόκληση για το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τις χώρες μέλη. Η ομάδα αυτή εργασίας, η ανοιχτή ομάδα ήταν μια ομάδα εργασίας κρατών μελών, τα έθνη είναι μέλος αυτήν την οργάνωση και εκεί ε, βασικά επικεντρώνομαι. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με μία φωνή και να μιλήσουμε με μία φωνή σε μία ομάδα όπου οι χώρες ε, μέλη μοιραζόντουσαν ευθύνε ε, με εξωενωσιακές χώρες μέλη. Πραγματικά ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα και θα πρέπει να πω ότι όλα πήγαν καλά. Δώσαμε συγχαρητήρια στον εαυτό μας. Ε, πραγματικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και δεν δημιουργήσαμε μια άλλη υπηρεσία. Ε, αν είχαμε καταλήξει σε μια κοινή θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα έβαζε μαζί την ομάδα των 27 σε μια κοινή θέση. Θα ακούσουμε βεβαίω και τον εκπρόσωπο τη Αφρικανική Ένωση που θα μιλήσει μετά από μένα και μία από τι ενδιαφέρουσε εμπειρίε για μένα κατά τη διάρκεια αυτή τη άξιση είναι οι διάφορε απόξει ε, που ήρθαν στην επιφάνεια ε, στην ομάδα αυτή. Υπήρχαν ε, μικρά νησιά, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αναδυόμενες οικονομίες κτλ. Και πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ πλοκή αύξηση ε, άσκηση και τα καταφέραμε τουλάχιστον αυτή είναι η ανάλυση που κάνουμε εμείς ότι καταλήξαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θέσαμε πάνω από 170 στόχους και όλα αυτά θα μας ε, κρατήσουν δραστήριους για αρκετό καιρό. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επισέλθουμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της συζήτηση. Ήταν σημαντικό για μας να ληφθούν υπόψη τρεις διαστάσεις της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, το περιβάλλον, η ανάπτυξη, τα κοινωνικά θέματα, όλα αυτά τα λάβαμε υπόψη μας, αλλά έχουμε, θέσαμε και στόχους για θέματα για την ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν και συζητήθηκαν και, άλλα θέματα όπως οι στόχοι 66. Ε, ε, Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη προβολή του κράτους δικαίου. Επετέχθη κάποια πρόοδος σε θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, αλλά σε ό,τι αφορά τον στόχο της διεθνούς εταιρικής σχέσης, έχουμε την αίσθηση ότι μερικοί από τους εταίρους μας βασίζουν την δουλειά που κάνουν σε μία μάλλον συντηρητική προσέγγιση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική βάση για τις εργασίες μας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της Δευτέρας Ιουνίου Χρησιμοποίησε λοιπόν αυτή τη βάση και εμείς θα πρέπει να στηριχτούμε εκεί για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα πριν ξεκινήσουν διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις. Γιατί όταν περάσουμε σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε πλέον να έχουμε την πολυτέλεια ε, περίεργων διαπραγματεύσεων στη διακυβερνητική διαδικασία θα πρέπει να μιλήσουμε με μία και μόνο φωνή χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές μεθόδους. Όπως γνωρίζετε, θα υπάρξει μια διάσκεψη κορυφής το Σεπτέμβριο του 2015 και οι λεπτομέρειες θα πρέπει να συμφωνηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή η συνάντηση των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων θα γίνει την τρίτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου του 2015. Βεβαίως επιμένουμε ότι η άποψη όλων των εμπλεκομένων του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συνυπολογιστεί και όπως ενδεχομένως γνωρίζετε από την εργασία των ΗΕ δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να προβληθούν αυτά τα επιχειρήματα γιατί δεν συμφωνούν όλοι με την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, δεν είναι τόσο ενθουσιώδης όσο εμείς. Το άλλο θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο η ύπαρξη της ανοιχτής ομάδας εργασίας. Υπήρξε ένα πάνελ υψηλού επίπεδου ε, το οποίο κατέληξε σε σημαντικό έργο και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να κάνει μια έκθεση σύνθεσης σχετικά με τα όσα συνέβησαν και αυτό θα πρέπει να υποβληθεί πριν από το τέλος της χρονιάς. Ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα MDGs. Ο Κόφι Ανάν έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο και είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό που κάναμε στην ανοιχτή ομάδα εργασίας να μην περιορίσει τη δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα να συμβάλλει. και να προδικάσει τις διαπαρβατεύσεις. Επίσης καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο πρόεδρος γενική έλευση. Είμαστε ευτυχείς που είναι Αφρικανός ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγάντα που ήταν πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης από το μέσο Σεπρεβρίου. Θα ετοιμάσει την όλη διαδικασία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα αναλάβει ένα άλλο PGA. Όλη η προπαρασκευαστική εργασία θα γίνει στην τέταρτη προπαρασκευαστική ε, συνεδρίαση. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, να υπάρξει ισορροπία των τριών αυτών διαστάσεων της ε, βιώσιμη ανάπτυξης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει, να συνυπολογιστεί και το κράτος δικαίου Διεξάγονται βεβαίως ακόμα μερικές συζητήσεις. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί τώρα. Μας απασχολεί η εισαγωγή ενός τέταρτου πυλώνα. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος, μου, πιέζει, ε, θα ήθελα να πω ότι το θέμα των κλιματικών αλλαγών είναι καθοριστική σημασία. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ένα θέμα ορατό, θα πρέπει όμως να μην υπάρχει, υπάρχει εμπλοκή με τη συνάντηση στο Παρίσι που βασικά έχει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Είναι καλό ότι θα πάρει το λόγο μετά από μένα εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης γιατί αυτό είναι ένα χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσε να διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γενικό Γραμματέας θεώρησε ότι η συμβολή μας είναι σημαντική, είναι συλλογική προσπάθεια όμως και θα πρέπει να συνεργαστούμε με άλλες περιφερειακές ομάδες και κυρίως με την Αφρικανική Ένωση που είναι ο μεγαλύτερος ετών θα λέγαμε ε, βιώσιμη ανάπτυξη λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζεται. Και θα θυμάστε όταν ε, έγινε η διάσκεψη κορυφή Αφρικανική Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, υπήρξε μια συμφωνία να συνεχίσουμε να συντονίζουμε τι θέσει μα και αυτό είναι κάτι που κάνουμε σε τακτική βάση πραγματικά θα μας δοθούν περισσότερες ευκαιρίες ε, να σκεφτούμε μια ευρύτερη ημερησία διάταξη, το θέμα της καταπολέμησης, της ένδυας, ε, το ρόλο της ε, κοινωνίας και αυτό θα το επιτύχουμε εάν η Ευρώπη και η Αφρική συνεργαστούν στο μέλλον. Και θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε ανυπομονησία να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επισκόπηση και τώρα περνάμε στον πρέσβη κύριο Τζάι Κουμαρ Μπράμντεο, πρέσβευτη της Αφρικανικής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλη, Αναπτύξεως που μου επιτρέπουν να έρθω για να εκθέσω την αφρικανική προσέγγιση στη συνεδρίασή σας. Κυρία Πρόεδρε η 22η τακτική σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ε, της Αφρικής Ενώσεως τον Ιανουάριο του 2014 υιοθέτησε τους στόχους για την ανάπτυξη στην Αφρική και κάλεσε την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης συνεργασία με τα κράτη-μέλη ε, να προχωρήσουν στην ενσωμάτωση στους υφιστάμενους ε, στις υφιστάμενους διαλόγους για την βιώσιμη ή αηφόρο ανάπτυξη στη διακυβερνητική ομάδα των στόχων αυτών, αλλά και στη Διακυβερνητική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αηφόρο χρηματοδότηση και την ατζέντα αναπτύξεως μετά το 2015. Με βάση τις αποφάσεις τον Απρίλιο του 2014 στην ε, Νέα Υόρκη υπευλήθησαν τα απαραίτητα εργαλεία στην ε, ομάδα της Νέας Υόρκης για την ε, ανάπτυξη από πλευράς αφρικανικής προσεγγίσεως για, την, για τον εμπλουτισμό της συστήσεως μετά το 2015. Οι έξι πυλώνες της κοινή αφρικανικής θέσεως και το σχέδιο στόχων δικτών και προσεγγίσεων συζητήθηκε διεξοδικά ώστε να είμαστε σίγουροι πως ευθυγραμμίζεται με τους στόχους αεφόρου ανάπτυξης. Συζητήθηκαν τα θέματα αυτά με τους πρέσβεις ε, στη Γενέβη και τις Βρυξέλλες τον, Ιούλιο του 2014 και εξετέθη εκεί η αιτιολογία και η στόχευση του κάθε στόχου, η διαδικασία διαπραγμάτευσης λοιπόν και τα προσεχή βήματα από το Σεπτέμβριο του 2015. Μένει να χαραχτούν. Μετά το 2015 λοιπόν η αφρικανική πλευρά ακολουθεί μια προσέγγιση αντίστοιχη με αυτή της Ατζέντας 2063. Μια 50 κονταετή δηλαδή προσπάθεια προγραμματισμού, ένα προγραμματισμό για 5 κονταετία, ώστε να είμαστε έτοιμοι για το 2063 από πλευράς Αφρικανικής Ενώσεως. Ξεκινήσαμε το 2013, όταν χαιρετήσαμε την 50η επέτειο της θεσπίσεως της, ε, του Οργανισμού Αφρικανικής Ενώσεως, που στη συνέχεια μετετράπησε Αφρικανική Ένωση. Έχουμε έξι πυλώνες στους οποίους εκτίθενται οι αποφάσεις μας με την αναδιάρθρωση της οικονομικής μεταρρύθμισης και ανάπτυξης, την τεχνολογία της επιστήμης και την καινοτομία, ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, περιβαλλοντικά αηφόρο ανάπτυξη, διαχείριση φυσικών πόρων, διαχείριση φυσικών καταστροφών ή κινδύνου φυσικών καταστροφών, ειρήνη και ασφάλεια και εν τέλει χρηματοδότηση και εταιρικές σχέσεις. Αυτή είναι οι έξι πυλώνες. 90% και άνω των κοινών προτεραιοτήτων ε, των Αφρικών θέσεων έχουν ενσωματωθεί σε αυτή την έκθεση, στην ομάδα. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές σε σχέση με τα πιο ε, λεπτά ζητήματα θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, διαφάνεια στη διακυβέρνηση, την παράνομη χρηματοδότηση και λοιπά ζητήματα. Η κύρια πρόκληση λοιπόν εδώ έχει να κάνει με τη βούληση για, εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Η επίτευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στα επιμέρους ζητήματα και κυρίως τους κινδύνους για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και ανάλογα βέβαια και με την προσέγγιση, τη στρατηγική που θα υιοθετηθεί για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Εν προκειμένου, προβλήματα που έχουν ε, εντοπιστεί στο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης ε, και κυρίως οικονομικής διαχείρισης που είδαμε, τη χρηματοπιστωτική κρίση, όλα αυτά αποτελούν διδάγματα για μας με τις συνέπειες που είχαν για τις κοινωνίες, τα άτομα, τις οικογένειες και επιβάλλονται σιγά σιγά πιο αυστηρές διατάξεις και επιτήρηση στους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να εμφανιστούν αντίστοιχα προβλήματα σύντομα. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις οικονομικής ε, διαχείρισης πάνω απ' όλα, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στις αφρικανικές χώρες. Προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου, είτε στην, ε, ε, ε, στην περιορισμένη ισχύ των θεσμών, στην ασθενή την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης ή την, τις επιλογέ επιλογές προσώπων, στα οποία βεβαίως μπορεί να έχουν επίδραση και διεφθαρμένα στοιχεία, πάνω στα οποία είναι οικοδομημένες μερικές φορές οι κοινωνίες. Με μια μεταρρυθμισμένη λοιπόν προσέγγιση και από τα Ηνωμένα Έθνη που μπορεί να προσφέρει συστημική ε, συνοχή στην παγκόσμια οικονομική διαχείριση και για καλύτερη διαχείριση των θεσμών και των αρχών μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια μεταρρύθμιση οικονομικών θεσμών που θα ενίσχυαν την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση στο ίδιο, την ίδια τοποθέτηση μπορούμε να υιοθετήσουμε και για την πολιτική διαχείριση. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο της πολιτικής διαχείρισης, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, πολύ χειρότερες από αυτό της οικονομικής διαχείρισης. Και το έχουμε δει στο παρελθόν, δυστυχώς, όταν ηγέτες ε, αιμοσταγείς ή ε, αδίστακτοι μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευση χώρες ολόκληρες. Πρέπει λοιπόν εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν το χρηστό δρόμο της διακυβέρνησης να ενθαρρυνθούν και να δουν ανταμοιβή ε, για τις προσπάθειές τους. Εκείνοι οι οποίοι έχουν επιλέξει τον δρόμο της δημοκρατίας και των ε, θεμητών ε, επιλογών δεν θα πρέπει να καταδικάζονται στη φτώχεια, στην, στον αποκλεισμό από την υγεία, τη την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον ηλεκτροδότη, την ίδρυυση, τα σχολεία και έτσι χρειάζεται στόχοι με σαφή προσέγγιση ανάπτυξης που θα επιτρέψουν σε όλους τους αρχηγούς κυβερνήσεων να αποδείξουν κιόλα ότι είναι λειτουργική η δημοκρατία. Και έτσι όλο, όλος ο πληθυσμός όπου είναι φτωχή, είτε πρόκειται για την Αφρική είτε πρόκειται για την Ευρώπη, θα πρέπει να εξασφαλίζει δυνατότητες για εκπαίδευση, για ανάπτυξη δεξιοτήτων και για προετοιμασία στην εμπλοκή στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να αποτρέψει την εμφάνιση φαινομένων ε, νεολαίας χωρίς προοπτικές, με τάσεις ακραίες, με τάσεις οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο και για την ειρήνη, αλλά και να οδηγήσουν πολύ σοβαρότερες συνέπειες. Άρα χρειάζεται υποστήριξη αυτών ακριβώς των κυβερνήσεων. Μέχρι τώρα η περιφερειακή ή διεθνής ή και διεθνής παρέμβαση είχε ανάμεικτα αποτελέσματα, κυρίως στην Αφρικανική Ήπειρο και την ανάπτυξή της. Οι βασικές αιτίες της αστάθειας και της οικονομικής ανέχειας πρέπει να καταπολεμηθούν, πάνω απ' όλα πρέπει να καταπολεμηθεί η ανέχεια προληπτικά αλλά και με επικοδομητικά μέτρα μέσω παραδείγματι της υιοθέτηση κανόνων ε, εμπορίου και επενδύσεων θεμητών, ισοδίκαιων, που να επιτρέπουν την ανάπτυξη όλων των χωρών. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ της αναπτυξιακής, του αναπτυξιακού θεματολογίου ή ατζέντα και της, ε, του θεματολογίου για την ανάπτυξη πλούτου ή ευημερίας. Αυτό το θεματολόγιο θα πρέπει να αντικαταστήσει την ανάπτυξη μεν, χωρίς όμως αυτή η μετάβαση να παραμελήσει πιθανές δυσμενείς συνέπειες από τη μετάβαση. Κακή πολιτική, οικονομική, δημοσιονομική διαχείριση έχει οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις στην Ήπειρό μας σε συγκρούσεις ένοπλες και ξέρετε ότι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα διαχείρισης ένοπλων σειράξεων ή επίλυσης κρίσεων πάρα πολύ συχνά. Είχαμε, όπως είπα, ανάμεκτα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις ε, της διεθνούς κοινότητας των περιφερειακών δυνάμεων. Ε, πολλές φορές μπόρεσαν να αποτρέψουν ε, προβλήματα, αλλά όχι πάντοτε και πολλές φορές τα αποτελέσματα ήταν πολύ δυσμενέστερα από την ίδια την ενόπλη κρίση. Πρέπει δηλαδή να είμαστε θέση να γνωρίζουμε πώς πρέπει να παρέμβουμε και σε ποιο βαθμό. Εκτρεμιστικές οργανώσεις οι οποίες αναλαμβάνουν τρομοκρατική δράση για να επιτύχουν τους στόχους τους έχουν οδηγήσει σε απίστευτη αθλειότητα εξαθλίωση και δεινά πολλά μέρη της Αφρικής και κυρίως την περιοχή του Σαχέλ. Η, η Αφρικανική Ένωση έχει στηρίξει τις προσπάθειες της Αφρικής για την εξασφάλιση της ε, ε, ειρήνης και της ευημερίας. Μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη η σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο. Η εταιρική αυτή σχέση λοιπόν και συνεργασία Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ επιτυχής ε, με το μεικτή ιδιαίτερα με την κοινή ιδιαίτερα στρατηγική Αφρικανικής Ανάπτυξης και για την διαχείριση και σχεδιασμό της αφρικανικής διακυβέρνησης και οικονομικής δράσεως. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο για να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η ευημερία. Κυρία Πρόεδρε, στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, οι ε, δυσμενείς επιπτώσεις και συνεπείς κλιματικής αλλαγής είναι ορατές σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αφρικανική Ήπειρο. Χρειάζεται λοιπόν να κινητοποιηθούν επαρκείς και προβλέψιμοι πόροι από τις χώρες που προσφέρουν υποστήριξη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο σχετικό ταμείο. Μέχρι το 2020 θα χρειαστούν πολύ ψηλά κονδύλια και ελπίζουμε στη συνεργασία μεταξύ Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με, τα, τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα χρειαστεί ένα σύστημα βεβαίω για να ανισχυθεί η διαχείριση του κινδύνου, η πρόβλεψη και η αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και να αναλυφθούν τα μέτρα εκείνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Χρειαζόμαστε την συμμετοχή όλων των κρατών, μικρών, νησιωτικών, εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο για, την, το μετριασμό των συνοπιών της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ιστορικά εταίρος σημαντικός, οικονομικός, πολιτικός, ε, και ανθρωπιστικός βέβαια και στην ανάπτυξη δεν μπορεί λοιπόν να παραγνωρίσει τις, ε, τη συμμετοχή της στην κλιματική αλλαγή, στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και για την Αφρική. Και κλείνοντας κυρία Πρόεδρε θα ήθελα πολύ σύντομα να στραφώ στην εφαρμογή της χρηματοδότησης και των εταιρικών σχέσεων που θα χρειαστούν εφόσον εφαρμοστούν οι, ε, οι βιώσιμοι στόχοι ανάπτυξης στην προσεχή περίοδο. Αυτό σημαίνει μια πολυεπίπεδη δράση σε διάφορους τομείς με ε, κινητοποίηση πολλών πόρων εσωτερικών, δράσεις που έχουν να κάνουν με τον μετριασμό των παράνομων χρηματοπιστωτικών ροών και την ενίσχυση των κινήτρων για την ανάπτυξη, αλλά που φτάνουν μέχρι την, ε, και τα φορολογικά κίνητρα. Χρειαζόμαστε καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης. Χρειαζόμαστε, χρειάζεται να κοιτάξουμε ποια είναι η πραγματικότητα των ε, και πού βρίσκονται τα κλαπέντα αγαθά, ε, περιουσιακά στοιχεία των Αφρικανικών κρατών, να κοιτάξουμε πώς θα γίνει η διαχείριση της χρηματοπιστωτικής ε, λειτουργίας, να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης, εταιρικών σχέσεων για το εμπόριο, ενίσχυση κατά 30% έως το 2030 του ενδοαφρικανικού εμπορίου Χρειαζόμαστε προαγωγή των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων και μεταφορά τεχνογνωσία στην Αφρική, που πιστεύουμε ότι θα ε, κριθεί απαραίτητη, και βέβαια διαχείριση των κοινών αγαθών της Ιφιλίου, αντιμετώπιση δηλαδή κλιματικής αλλαγής, επιδημιών, παγκόσμια ε, αρχιτεκτονική και συνέπειες ε, ή συμπεράσματα καλύτερα από τον τελευταίο γύρο της Δόχα. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι έχω εξατλήσει το χρόνο μου και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο, μόνο, δύο ακόμα ομιλητές που εκπροσωπούν ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον, ε, τα Ηνωμένα Έθνη ε, και αυτοί θα πάρουν το λόγο μετά. Οπότε, το πολύ 20 λεπτά για ερωτήσεις, αν χρειαστεί, ενδεχομένως να μην γίνουν ερωτήσεις. Μήπως μπορείτε να μείνετε μέχρι το τέλος. Εσείς πρέπει να φύγετε. Α, ο ένας από τους ομιλητές θα πρέπει να φύγει, οπότε ε, να επανέλθουμε, ε, να κάνουμε ερωτήσεις τώρα και μετά να επανέλθουμε για περισσότερο. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Στίερ και ο κύριος Βάρινεν προς το παρόν. Τρεις ερωτήσεις λοιπόν. Θα τις πάρουμε και μετά θα περάσουμε στην επόμενη συνεδρία. Ε, κύριος Γκέρενς, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η δική μου παρατήρηση έχει πολιτικό καθαρά χαρακτήρα. Έχουμε μπροστά μας δύο μιλητές, οι οποίοι μας έδωσαν μια παρουσίαση για την κατάσταση και τη βάση πάνω στην οποία θα μπορούσαν να επιτύχουν οι διαπραγματεύσει. Δεν βλέπω καμία απόκληση μεταξύ του. Δεν διαπιστώνω την παραμικρή απόκληση και αυτό το διατυπώνω ω φοροτιμή στον τρόπο με τον οποίο εξέθεσαν το πρόβλημα. Νομίζω ότι μπορούμε αυτό το θεωρήσουμε ω καλό ιονό για μια διαδικασία η οποία ξεκινάει αλλά προ... Ε, προβλέπεται δύσκολη. Μια σύγκληση στις τοποθετήσεις στην Τόχα είχαμε διαπιστώσει και πριν από 10 χρόνια και όμως στο τέλος οι διαπραγματεύσεις κατέρευσαν, απέτυχαν. Διαπραγματεύσεις που είχαν να κάνουν με άλλο θέμα, το οποίο όμως πάλι άμεσα συνδέεται με το σημερινό μας ε, θέμα συζήτηση και που όμως με έκπληξη διαπιστώσαμε η 90 20, G110, ήταν εκείνη η οποία οδήγησαν σε αποτυχία τη συμφωνία. Δεν θέλουμε λοιπόν να επαναληφθεί αυτό. Γι' αυτό παρακαλώ ε, να μου απαντήσουν ο εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης αλλά και εκείνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξής ερώτηση. Διαθέτετε τα μέσα να ενώσετε τις προσπάθειες αφού μεταξύ σας δεν διαπιστώνετε διαφορά, ώστε να εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα εκείνη η οποία στο τέλος της δικασίας θα επιτρέψει να μετακινηθούν κάποιες κόκκινες γραμμές. Βλέπετε δηλαδή μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης βεβαίως και με τους άλλους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα θέματα της ανάπτυξης, διότι βλέπω ότι είμαστε πιο κοντά εμείς στις, ε, στην αντιμετώπιση, στην απάντηση στις ανησυχίες των Αφρικανικών κρατών. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να κάνουμε αυτό το επιπλέον βήμα και να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία θα αναπτυχθεί με κοινέ δυνάμεις, με κοινά μέσα. Είστε διατεθειμένοι να προβείτε σε αυτό το επιπλέον βήμα. Είναι πολύ σημαντικό και επιπλέον διαπιστώνω και από τις τελευταίες συζητήσεις ότι πάντοτε εμείς την ευηκονούς στους ε, εταίρους, ότι η εταιρική σχέση όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε αποτελεί μια καλή βάση συζήτησης και ότι μπορεί να έχετε και άλλους εταίρους μεν, αλλά δεν τίνουν το ίδιο, το ίδιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματά σας. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ Εάν αυτή η λογική, αυτή η στρατηγική για τη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο αυτών ε, ενώσεων, ομάδων κρατών, Αφρικανικής και Ευρωπαϊκής, είναι δυνατή. Ευχαριστώ κύριο Στίερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίζω την ε, ευκαιρία που δίνεται για συζήτηση αυτή την πρώιμη ε, φάση που μπορεί να έχει και διδακτικό θα έλεγα χαρακτήρα ως προς την ανάπτυξη των σχέσεων και μια κοινή θέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης για, την, ε, για το θεματολόγιο μετά το 2020. Έχουμε πολύ πλούσια εμπειρία από τις εργασίες της ομάδας εργασίας, τους στόχους. Ο κύριος Πρέσβης άλλωστε κατέστη σαφές και ήταν πολύ ενδιαφέρον το τι, δουλειά, το τι δουλειά γίνεται για το συντονισμό των θέσεων. Ε, ένα ή δύο σημεία θα έλεγα είναι πολύ σημαντικά. Αναφερθήκατε στις ε, προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια το άρθρο 16 και τη σημασία που αποδίδεται στο κράτος δικαίου και την τήρηση των κανονών του κράτους δικαίου, όπου δυστυχώς οι επιδόσεις δεν είναι ικανοποιητικέ και ελπίζουμε ότι θα ενταχθεί το θέμα αυτό στη συζήτηση και ότι θα ενισχυθεί η σημασία του. Ρωτώ όμως, εάν διαβλέπετε κάποιες πιθανές συμμαχίες προκειμένου να φτάσετε σε καλύτερα επίπεδα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάρινεν. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαίρετης παρουσίαση και αποτελούν πολύτιμη βάση αξιολόγηση όταν αρχίσουμε να διατυπώνουμε την έκθεσή μας για την αξιολόγηση του θεματολογίου μετά το 2015 όπου πιστεύω ότι να ξεκινήσουμε το χειτερό δυνατό. Ε, κοιτάω λοιπόν την έκθεση που πήρα για πρώτη φορά στα χέρια μου σήμερα και δεν ξέρω γιατί και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαπιστώνω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο πολύ επικίνδυνο, ότι δηλαδή διατυπώνονται υπερβολικά υψηλό αριθμό προτεραιοτήτων. Έχουμε υπερβολικά πολλέ προτεραιότητε και χρειάζεται ω εκ τούτου μια διάρθρωση στου συλλογισμού μα, στο σχεδιασμό μα, στη διατύπωση των εκθέσεων και των εγγράφων όπω αυτά εδώ. Έχουμε δύο κύριου στόχου. Περιορισμό τη φτώχεια και προαγωγή τη αηφόρου ανάπτυξη. Πολλά από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σαν στόχους είναι περισσότερο μέσα για την επιτεύξη αυτών των δύο στόχων. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούμε εγκάρσια να παρακολουθήσουμε και να υποστηρίξουμε σε κάθε αναπτυξιακή πολιτική. Ερωτώ λοιπόν και διαρωτώ με, εάν στη δική σας δουλειά και, στα και στην ε, Νέα Υόρκη έχετε χειριστεί, έχετε δει τα ζητήματα αυτά και το ενδεχόμενο ομαδοποίησης ώστε να περιοριστεί αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός στόχων μέσων προτεραιοτήτων που καταγράφονται στον τομέα αυτών. Έχω και εγώ ετοιμάσει ένα σύντομο έγγραφο ως βάση συζήτησης, ε, το οποίο θα ήθελα να διανύμω και στους συναδέλφους της Επιτροπής, ώστε να δούμε εάν με βάση αυτό μπορούμε στην έκθεσή μας να ε, συμβάλλουμε με κάποια, κάποιο συγύρισμα, κάποια υποστηρή τάξη και διαβάθμιση μεταξύ προτεραιοτήτων και μέσων, εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Αλλά ρωτώ ποια είναι η δική σας εμπειρία και αν έχετε κάποιες ε, ιδέες ήδη για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό στη διαδικασία. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ο κύριος Μάρτιν Πάρτ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύκο, αν δεν απατώμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος Ο Πρέσβης εξήγησε πολύ καλά την κατάσταση στα, στη Νέα Υόρκη. Το Σεπτέμβριο του 2015 θα πρέπει, όπως προχωρούμε στη διαδικασία αυτή, να έχουμε υπόψη δύο στοιχεία. Καταρχάς, ποια είναι τα αποτελέσματα των προσπαθειών για ένα θεματολόγιο οικουμενικό, που δεν πρέπει να λησμονηθεί, και επίσης το ότι το θεματολόγιο θα πρέπει να εξισορροπεί τους στόχους που είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και η ενίσχυση της ε, αηφόρου ανάπτυξης ως κυρίους στόχους, ως ε, πρωταρχικούς στόχους. Εξέθεσε ο πρέσβης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαδικασία του προσδορισμού των στόχων, αλλά για τα αποτελέσματα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε μια καλή βάση για να προωθηθούν οι στόχοι, χωρίς να είναι τέλεια. Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω ότι καταγράφονται στο έγγραφο πορισμάτων. Συμφωνώ με τους λοιπούς ομιλητές ότι ίσως είναι υπερβολικά πολλοί οι στόχοι και Ίσως χρειάζεται μια ομαδοποίηση, καλύτερη ίσως καταγραφή των ε, συσχετισμών, ώστε να γίνουν πολιτικά πιο ελκυστικά, αλλά και εύληπτα τα πορίσματα αυτά και οι στόχοι. Στους προσεχείς μήνες ε, πολλές από τις προσπαθίες μας θα εντοπίσουν ε, κυρίως μέσα εφαρμογής και είχαμε επίσης μια πολύ καλή έκθεση της ομάδας ε, πραγματογνωμόνων για τη χρηματοδότηση της αηφόρου ανάπτυξης. Έκθεση η οποία καταγράφει τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτεραιότητες της κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό. Αποτελεί όμως μια μόνο αρχή στη διαδικασία αυτή. Χρειάζεται μια άλλη, μια άλλη υπουργική διάσκεψη τον ε, Ιούλιο στην Αντισαμπέμπα για να προετοιμαστεί η διάσκεψη αυτή που θα αποτελέσει τη συνέχεια της ε, διάσκεψης του Μοντερέι. Θα είναι περιπλοκή. Ε, περίπλοκα τα θέματα των συζητήσεων και οι εργασίες και με χαρά ακούω από τον πρέσβη Μπραντέο ε, να διατυπώνεται έκθεση, ε, έμφαση ως προς την κινητοποίηση των πόρων γιατί θα είναι πολύ φιλόδοξο το θεματολόγιο πιστεύω και θα πρέπει για το λόγο αυτό στη συζήτηση να διατεθούν όλα τα μέσα, να μπουν όλα τα μέσα εφαρμογής που είναι διαθέσιμα. Μικρό στοιχείο μόνο είναι χρηματοδότηση, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει όλο και περισσότερη συμφωνία στη Νέα Υόρκη και συνένεση ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν ε, ε, εθνικοί πόροι και εθνικές πολιτικές να αναπτυχθούν. Αυτά λοιπόν πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ, σημαντικές, ε, πολύ σημαντική απόδοση των προσπαθειών το Σεπτέμβριο του 2015 με την ολοκλήρωση της Βεβαίως και προσβλέπουμε στην ε, υποβολή της έκθεσης της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχετε ανακοινώσει το τέλος του έτους. Χρειάζεται να δούμε την έκθεση, χρειαζόμαστε ουσιαστικά συμπεράσματα το Δεκέμβριο για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μια ε, στεναρή ευρωπαϊκή θέση, μια ρωμαλαία ευρωπαϊκή θέση για τις διαπραγματεύσεις. Περιμένουμε λοιπόν την έκθεσή σας και για τους ε, βουλευτές αλλά και για τον πρέσβη Μπραντέο θα ήθελα να αναφερθώ στην θέση της Αφρικανικής Ένωσης, στην Κοινή Αφρικανική Ένωση, η οποία είναι ένα αξιόλογο επίτευγμα, σημαντική συμβολή στη διαδικασία και επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι πιστεύουμε, όπως άλλωστε είπε και ο κύριος Γκόρενς ότι προσεγγίζει σημαντικά, ο κύριος Γκόρενς ότι προσεγγίζει σημαντικά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Ξεκινήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της ε, διασκέψεως, την προετοιμασία της ε, διασκέψεως, η οποία μας έδωσε εντολή να συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης. Είμαστε στη διάθεση της Αφρικανικής Ένωσης εφόσον επιθυμεί να ξαναρχίσει ο διάλογος των ταχύτερο δυνατόν διότι πιστεύουμε όπως και οι άλλοι ομιλητές, ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική είναι σε θέση να διατυπώσουν κοινή τοποθέτηση, κοινέ θέσει και από τον Ιούνιο του 2014 και την Αφρικανική ε, κοινή διακήρυξη νομίζω ότι είναι σαφές πως έχουμε σαφές το περιθώριο για κοινέ θέσεις και ως εκ τούτου θα ήθελα να πω ότι προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτού του ε, διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους μας. Επιτρέψτε μου να κάνω μία ερώτηση. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για τη διαδικασία εν ώψη συμφωνίας. Αν θέλουμε να ε, λειτουργήσει αυτό, θέλουμε και πολιτική υποστήριξη. Μιλήσατε για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε όχι μόνο στο πώς, αλλά και στο γιατί κάνουμε αυτό ε, που κάνουμε, τι έγινε την προηγούμενη φορά, τι επιτεύχθη την προηγούμενη φορά, ε, τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για την επόμενη φορά. Και έτσι θα συμφωνήσει μαζί μας και εκείνη η γνώμη. Δηλαδή, αν ο κόσμος κληθεί να προσέξει, να πληρώσει, θα πρέπει να ξέρει για ποιο λόγο. Πρέπει να ε, δώσουμε επιχειρήματα, να πείσουμε την κοινή γνώμη ε, και στις ανεπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες για να λειτουργήσει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε πέντε λεπτά ο καθένας το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κατα... Ξεκινώντας με... από τη δική σας ερώτηση, ε, λυπάμαι που απαντώ σε μια ουσιαστική ερώτηση μιλώντας για τη διαδικασία και πάλι. Αλλά πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ε, εν γέννη γνωστό, είναι ο ισχυρότερος υποστηρικτής των δικαιωμάτων της κοινωνίας των πολιτών ε, και υπάρχουν προβλήματα με κάποιους άλλους τα Ηνωμένα Έθνη. Και νομίζω ότι μια απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ακουστεί φωνή, η κοινωνία των, να ακουστεί η κοινωνία των πολιτών και το κοινοβούλιο. Και βεβαίως η, της χιλιετίας ε, προέκυψαν από μια τέτοια διαδικασία. Και όταν μιλάμε για κοινωνικά ζητήματα αυτό είναι σημαντικό ε, ακόμα περισσότερο. Θα πω επίσης, μιλώντας γαλλικά λέει ο Πρόεδρος, ε, ε, σε απάντηση τον κύριο Λόρενς, όπως και τον κύριο Μάρτιν Πράντα με τον οποίο είχαμε εξαιρετική συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι οι θέσεις μας πολύ κοντά. αν δείτε τις λεπτομέρειες του εγγράφου θα διαπιστώσετε κάποια σημεία που υπάρχουν διαφορές από τη μία την άλλη πλευρά. Πρέπει επίσης να πούμε ότι όταν ε, βρισκόμασταν ακόμα στο Ρίο για τη διαδικασία Ρίο Ρίο-Συνήκωση υπήρχε στενότατη συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές και θα θυμόσαστε ίσως οι δύο πλευρές ήταν υπέρ ε, τη, μιας νέα, ενός νέου διεθνού οργανισμού για το περιβάλλον με έδρα την Αφρική. Εξ όσων ε, αντιληφθήκαμε αυτό δεν κατέστη δυνατόν τότε, δεν φταίμε ε, και λόγω ημών αλλά και λόγω των Αφρικανών φίλων. Παρά τα αυτά παραμένει σημαντικό, μπορώ να μιλήσω ε, ανοιχτά. Είναι σημαντικό οι Αφρικανοί φίλοι μας να καταφέρουν να επιβάλλουν τη θέση τους στο πλαίσιο των G77. Και όπως είπατε είναι ετερογενής ε, ομάδα μερικές φορές, αλλά ε, στο εσωτερικό αυτής της ομάδας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αφρικανοί φίλοι μας είναι οι πιο κοντινοί εταίροι μας. Επίσης αυτό ισχύει ότι αν προέρχεται κανείς από, από ένα μικρό νησί του Ειρηνικού θα διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση επειρασπίζεται πιο πολύ τα συμφέροντά σας στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με τους ε, άλλους εταίρους σας οι οποίοι είναι τεχνική συμμαχοί σας ε, στις, ε, στον διαπραγματεύτο του ΟΗΤΕ. Πρέπει όμως να ενισχυθεί και να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία γιατί πολύ περισσότερα θα γίνουν στη Νέα Υόρκη. Έχουμε εξαιρετική επαφή με, την, με τους Αφρικανούς εταίρους μας, την αντιπροσωπεία της Αφρικανικής Ένωσης και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε Επίσης θα πω δύο λόγια και μιλά αγγλικά ο μιλητής ε, για το λεγόμενο clustering, την ε, ε, δημιουργία ομάδων. Ο Κόφι Ανάν το έθεσε το θέμα και είχε την αρχή να διατυπώσει ένα σύντομο κατάλογο στόχων της χιλιετίας. Δεν θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά αν δεν είχε παρέμβει. Εν μέρη λοιπόν επειδή υπάρχει η προσέγγιση του Φκόφια ε, Ανάνο που ήταν σπουδαίος Αφρικανός και γενικός γραμματέας δεν ήταν ε, ε, τόσο δημοφιλής ε, στο Νότο όσο ήταν σε εμά, υπάρχει το αίσθημα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεύτερη φορά. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η διακυβερνητική διαδικασία τη ανοιχτή ομάδα εργασία και εξακολουθεί να χρειάζεται κάποια ε, προσπάθεια για να, για να διατηρηθεί αυτή η προσπάθεια του ε, Γενικού Γραμματέα. Εν πάση περιπτώσει, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνο να ακολουθήσουμε το δρόμο της ε, προσέγγισης του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Όλοι έχουν κάτι που είναι σημαντικό για αυτούς και θέλουν να το προσθέσουν στον κατάλογο. Το γεγονός ότι ο κατάλογος είναι και αρκετά, η κατάσταση είναι αρκετά καλή, η, οφείλεται και επίσης και στο γεγονός ότι συμπρόεδρος, συμπρόεδροι ήταν ε, ένας Ευρωπαίος και ένας Αφρικανός, ο, οι πρέσβεις της Ουγγαρίας και της Κένια που ε, λειτουργήσαν εξαιρετικά. Τώρα, το θέμα της ομαδοποίησης Τη της συνάφρησης, της μείωσης του αριθμού των θεμάτων. Ε, και πραγματικά πρέπει να πω ότι θα υπήρχε κίνδυνος. Αν αρχίζαν να περι, οι περικοπές, δεν θα, ήταν, ε, δεν θα ανάγκη, κατά ανάγκη αυτά που θεωρούσαμε εμείς περιτά, αλλά ενδεχομένως αυτά που αφορούν τη σωστή διακυβέρνηση, την, το κράτος δικαίου και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Έτσι, από τη στιγμή που αρχίσει κανείς να κάνει περικοπές, <laughs> πρέπει να φροντίσει ότι δεν θα περικοπούν ε, τα, αυτά που δεν θέλουμε να φύγουν από τον κατάλογο. Και επίσης πρέπει να πω ότι ε, ε, ε, αν στραφούμε προς το Γενικό Γραμματέα και αυτός κάνει μια σύνθεση θα, το, θα κάνει κάποιες περικοπές. Εγώ δεν, θα, δεν περιμένω θαύματα στον τομέα αυτό. Είναι πιο σημαντικό όταν μιλάμε για τον κάθε στόχο να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν και ένα από τα θέματα έχει σχέση με το ότι πρέπει να επιμείνουμε να, έχουν, να είναι ε, στόχοι με νόημα, να έχουν ουσία. Πρέπει να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια, αλλά αν μου ζητήσετε να, να πω εγώ τι πιστεύω ότι θα γίνει, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε δισέλιδο. Θα είναι κάπως ε, ε, βαρβαρημένος ο κατάλογος να δούμε τι θα πάρουμε και πάντως εμείς θα προσπαθήσουμε ε, να προχωρήσουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πω ότι πρέπει να επανέλθουμε για κάποια θέματα που δεν πετύχαμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλαμε. Θέλαμε το κράτος δικαίου να είναι σε ε, σημαντικότερη θέση και πιστεύω ότι έχουμε τέρους σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι σημαντικό όπως στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, να μην ε, κάνουμε το θέμα αυτό ε, ένα θέμα αντιπαράθεσης βορρά-νότου ή ανατολής-δύσης. Αν επιμείνω στο θέμα της ε, ένομης τάξης, του κράτους δικαίου, η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ένα σημαντικό ζήτημα και αυτό έχει σημασία γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δουλέψει πολύ από αυτού. Όταν μιλάω για αυτά τα θέματα είναι απολύτως σαφές ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κανόνες σε άλλες περιοχές του κρατους δικαιου η αντιμετωπιση της διαφθορας ειναι ενα σημαντικο ζητημα και αυτο εχει σημασια γιατι το ευρωπαικο κοινοβουλιο εχει δουλεψει πολυ απο αυτό. οταν μιλαω για αυτα τα θεματα ειναι απολυτως σαφες οτι δεν θελουμε να επιβαλλουμε κανονες σε αλλες περιοχες του κοσμου πράγματα τα οποία εμείς δεν θέλουμε να αποδεχτούμε. Γιατί αυτό που δεν είπα τώρα σε σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και τους αναπτυξιακούς στόχους χιλιετίας είναι ότι οι δεύτεροι ισχύουν για όλους, εφαρμόζονται για όλους συμπεριλαμβανομένων και ημών. Και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό πρέπει να, να συνεχίσουμε με τη μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένης, αν μου επιτρέπετε να πω, και τη διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης της δημιουργία, ισχυρή διαπραγματευτικής σχέση, γιατί χρειαζόμαστε να καταλήξουμε σε κάτι, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ευχαριστώ τον Πρέσβη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με την παρέμβαση του πρέσβη Χάρτινγκ. Θα ήθελα απλά και μόνο να προσθέσω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης και από τη στιγμή που του δίνουμε τη βαρύτητα που αξίζει ο διάλογος θα φτάσει σε ένα σημείο που θα μας οδηγήσει στο να υιοθετήσουμε και νέες θέσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο διαφόρων φορέων. Το σημαντικό είναι να επιτυχάνετε κριτική μάζα. Μπορεί και να μην συμφωνούμε πάντοτε σε όλα τα θέματα, αλλά πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τα περισσότερα θέματα, αν ο τρόπο σκέψη μα είναι παρεμφερή, δίχω άλλο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την κριτική μάζα. Υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες και έχουν παρατεθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν όμως θέματα που αφορούν και τους μεν και τους δε. Εάν τα αντιμετωπίσουμε αυτά εξετάζοντας τη σχέση αιτίου και αιτιατού αυτό δίχως άλλο θα μας επιτρέψει να επιδεντρώσουμε την προσοχή μας στις βασικές δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν και που θα πρέπει να έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Γιατί μας απασχολεί το τι συμβεί μετά το 2015. Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή οι άνθρωποι να μπορέσουν να αγγίξουν την ανάπτυξη. Για πάρα πολύ χρόνο Ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ε, αναζητούσαν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, προσέβλεπαν σε αυτό. Και ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους ακόμα και στα κατώτερα επίπεδα, καθώς και τα μέτρα που θα υιοθετηθούν, δίχως άλλο θα επηρεάσουν θετικά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τους δύο πρώτους ομιλητές για την ανασκόπηση που έκαναν. Περνάμε τώρα στο επόμενο πάνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον πρέσβη κύριο Χάτινγκ. Ωραία. Ακούσαμε τα όσα είχαν να μας πούν οι δύο πρέσβεις, οι οποίοι εργάζονται σε επίσημο επίπεδο. Τώρα έχουμε δύο ακόμα ομιλητές. Πρώτος είναι ο Σέμους Τζέπερσον, διευθυντής του Concord. Το Concord είναι μια πάρα πολύ σημαντική οργάνωση, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΜΚΟ ε, που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης. Δηλαδή συγκεντρώνονται όλες οι βασικές ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα ανάπτυξης. Ελπίζω ο κύριος Τζέφερσον θα έχει να μας πει πολλά και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Όλε Λούντ Κάνσεν, επικεφαλής της πλατφόρμας LED του Παγκόσμιου Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επειδή θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας το ρόλο του ιδιωτικού τομέα, η παρέμβαση του κ. Χάνσεν θα πάρα πολύ σημαντική. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα δοθεί πρωτεύον ρόλο στους χώρους πόρους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει βεβαίως να λάβετε υπόψη σας τα όσα είπαν οι δύο προλαλήσαντες ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πλούτου και ανάπτυξης. Καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι οι ομιλητές έχουν 10 λεπτά ο καθένας στη διάθεσή του. Ο κύριος Τζέφερσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια για το Concord. Το όνομά μου είναι Τζέφερσον, είμαι διευθυντής του Concord το Concord είναι μια ευρωπαϊκή οργάνωση ΜΚΟ και εκπροσωπούμε ΜΚΟ σε δύο επίπεδα σε κάθε χώρα μέλος υπάρχει μια πλατφόρμα αναπτυξιακών ε, ΜΚΟ και αντιπροσωπεύουμε και την οικογένεια των μεγάλων ΜΚΟ, ε, Handicap International, Save the Children κτλ. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ, ε, είμαστε ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικοί. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαμε ο βασικός συνομιλητής για θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε στην Επιτροπή ε, Ανάπτυξης της σχέσης μας. Το παρελθόν ήταν πάρα πολύ καλή, την προηγούμενη φορενιά είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία και με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να συνεργαστούμε μαζί σας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, νέων προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας απασχολεί μια σειρά από θέματα το θέμα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη. Μας απασχολούν επίσης θέματα που αφορούν τη συνοχή άλλων πολιτικών που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Επίσης, μερικοί από εσά γνωρίζετε ότι η επόμενη χρονιά είναι το έτος ανάπτυξης και θα συνεργαστούμε ιδιαίτερα με την κοινωνία, με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα να μου επιτρέπετε να αναφερθώ σε τρεις πτυχές της, του χρονοδιαγράμματος μετά το 2015. Το πρώτο είναι γιατί εμείς στην κοινότητα των ΜΚΟ θεωρούμε ότι αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία. Θα ήθελα να σας πω ποιε είναι οι απόψει μας για τα, ε, την εργασία της ε, Ανοιχτή ομάδα εργασία και να σας πω δύο λόγια σχετικά με το πώς βλέπουν τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης. Πιστεύω, όπως ανέφεραν ορισμένοι από τους ομιλητές, αυτό το πλαίσιο μετά το 2015, οι στόχοι δηλαδή βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία για μα, για τη γενιά μα. Καταγράψαμε ιδιαίτερη πρόοδο σε αναπτυξιακά θέματα, κρυζώσαμε την ακραία φτώχεια, αλλά βρισκόμαστε επίσης αντιμέτωποι ακόμα με βασικές προκλήσεις. Υπάρχουν ανισότητα, υπάρχουν, υπάρχουν θύλακοι ένδυας, υπάρχουν άνθρωποι που τους αφήνουν ανέγκυκτους ε, οι εξελίξεις. Ε, υπάρχει, ε, υπάρχουν κρίσεις, υπάρχει κλιματική αλλαγή που θα επηρεάσει και θα πλήξει τους πλέον ευάλωτους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνέχιση της ανάπτυξης με βάση μια λογική των, τη λογική των στόχων της χιλιετίας είναι κάτι καλό. Αυτό όμως από μόνο του δεν θα καταφέρει να επιλύσει το πρόβλημα, δεν θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Με άλλα λόγια, το να κάνουμε τα πράγματα με τον τρόπο που τα κάναμε στο παρελθόν δεν θα μας οδηγήσει εκεί που αποσκοπούμε να φτάσουμε. Αυτό δεν είναι μια δυνατότητα, μια επιλογή που έχουμε. Τι θα λέγατε αν μαθαίναμε από τους στόχους της χιλιετίας. Υπάρχουν διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε από τις επιτυχείς και ανεπιτυχείς προσπάθειες και όταν ε, οι προσπάθειε ε, δεν στέφτηκαν από επιτυχία θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Θα πρέπει να μιλήσουμε με μεγαλύτερη μεσότητα... σε όσου πλήττονται από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια παγκόσμια συζήτηση με όλου ε, του εμπλεκόμενου και θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι τι ακριβώ εννοούμε με τον όρο ανάπτυξη. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε συγκεντρώνοντα και νομίζω ότι το κάναμε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Θα πρέπει να μην εστιαστούμε μόνο στα συμπτώματα αλλά στις, στα αίτια και να συμπεριλάβουμε τις ε, αναντιστοιχίες των πολιτικών μας και ε, πάρα πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν σε μία παγκόσμια προσέγγιση. Το θέμα δεν είναι εμείς και εκείνοι. Το θέμα είμαστε εμείς σε αυτό το πλανήτη. Τέλος, κοιτάζοντας, εξετάζοντας το θέμα της ένδυας που ξεπερνάει το θέμα του εισοδήματο και εστιάζεται σε μια γενικότερη επιμερία των ανθρώπων. Όπως ανέφεραν οι ομιλητές, η διαδικασία της ανοιχτής ομάδας εργασίας ήταν μοναδική. Ε, κατέληξε σε συγκεκριμένους βιώσιμους στόχους, εμείς θα λέγαμε ότι συμφωνούμε με όλα όσα έγιναν και πραγματικά θα ενθαρρύναμε τη συνέχιση των διαδικασιών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μία βάση, δεν είναι ο απότερος ο στόχος ε, ξέρουμε τα συμπεράσματα των ε, ανοιχτών ομάδων εργασία, μπορείτε να τα διαβάσετε και εσεί. Θα ήθελα όμω να επικεντρωθώ σε τρία θέματα που μα δείχνουν πού θα πρέπει να επιτευχθεί κάποια βελτίωση. Ο πρώτος στόχος αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρονται στην εισαγωγή της έκθεσης, στο προήμιο της έκθεσης, αλλά δεν είδαμε μία προσέγγιση να διαπνέεται από ένα συγκεκριμένο ανθρωπιστικό πνεύμα και πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να διαχέεται παντού. Είναι βασικό στόχος που αφορά τη συμμετοχή των ανθρώπων που θα επηρεαστούν από τις πολιτικές και από τους στόχους. Και ε, να εξετάσουμε και το ρόλο που θα έχουν σε ό,τι αφορά αυτούς τους στόχους, την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το θέμα είναι αν θα συνεχίσουμε έτσι ή αν θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά το θέμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων πραγματικά μας βρίσκει σύμφωνος ο συγκεκριμένο στόχο, πιστεύουμε ότι είναι καθοριστική σημασία, θα επιθυμούσαμε να γίνουν περισσότερα και να καταλάβουμε πώς αυτό θα εφαρμοστεί. Πραγματικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε να ε, ασχοληθούμε με τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές και να επιτύχουμε την ισότητα. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν τομείς απασχόλησης, ε, και τον έλεγχο των γυναικών για διάφορα θέματα. Ε, αυτό απλά και μόνο σαν αφορά. Ένας τρίτος τομέας είναι η βιωσιμότητα στο περιβάλλον. Η εργασία, το έργο που επιτέλεσε η ανοιχτή ομάδα εργασία, άφησε ανοιχτό το θέμα αυτό των παγκόσμιων συνόρων. Δεν μπορούμε, των ορίων του πλανήτη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την τροχιά ανάπτυξη για πάντα. Υπάρχουν όρια στον πλανήτη μα. και στι διαπραγματεύσει θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευθύτητα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και καθώ και συγκεκριμένε προτάσει για το πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να πω ένα-δύο πράγματα. Πραγματικά μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο, αρμο... ο Επίτροπος Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συνεργάζονται προς την επίτευξη των στόχων. Και εγώ θα έλεγα στις ακροάσεις των επιτρόπων να θέσετε συγκεκριμένα ερωτήματα, να δείτε αν έχουν επιτευθεί οι στόχοι από πλευράς των επιτρόπων. Επίσης είχαμε πολύ καλή πρόσβαση στην Επιτροπή, στην χάραξη πολιτικών. Πραγματικά μας βρίσκουν σύμφωνους πολλά από αυτά τα θέματα. Σε ό,τι Βέβαια ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Είπατε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της άποψης ε, των διαφόρων απόψεων. Ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρική. Υπάρχει το θέμα της παγκοσμιότητας. Τι σημαίνει παγκοσμιότητα. Σημαίνει ότι θέτουμε ένα πλαίσιο ε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ποιος πληρώνει. Αυτό δεν είναι αξιόπιστο. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε παγκόσμιους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσει σε διαπραγματεύσεις και να αναλάβει δεσμεύσεις για τις ε, εγχώριες πολιτικές της. Ε, τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πιστεύω λοιπόν ότι στο πνεύμα της συνοχής θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή και τους συναδέλφους ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσουν τις πολιτικές που επηρεάζουν την ανάπτυξη σε άλλα μέρη του κόσμου. Ε, μιλήσαμε με τους εταίρους μας στο Μεξικό και μα, μας είπαν ότι εμείς δεν λαμβάνουμε πλέον ε, ενίσχυση από την ε, ε διμερή ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά και τις άλλες πολιτικές. Θα ήθελα να τελειώσω την παρέμβασή μου θέτοντας ένα άλλο θέμα. Την ανάγκη δηλαδή για δημιουργία, για αύξηση της ευαισθητοποίησης ε, του κοινού. Πιστεύω ότι οι τεχνοκράτες κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν ε, καλά. Εσείς κάνετε καλά τη δουλειά σας, αλλά χρειάζεται η κοινή γνώμη να γνωρίζει για τι πράγμα μιλάμε και για ποιο λόγο προτείνουμε τα όσα προτείνουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Ε, Χαίρομαι που είτε ο γιατί το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας μηχανισμός που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, θα ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Αυτό πέρα από τα ΜΚΟ, πέρα από την, ε, τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη. Υπάρχουν άλλοι τομείς για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό για μας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Um, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που μας υπενθυμίζετε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο, που ήδη διδραματίζει πιέζοντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. περνώ στον ε, δεύτερο ομιλητή, κύριο Λούντ Χάνσεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω να σας μιλήσω με τιμά πολύ. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την πλατφόρμα LEAD, η οποία ασχολείται κυρίως με τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στις Βρυξέλλες, αλλά και στην εφαρμογή των στόχων, των αναπτυξιακών στόχων. Θα σας δώσω με τις διαφάνειες που έχω φέρει κάποια στοιχεία πιο συγκεκριμένα, αλλά για να είμαι πολύ σύντομο, το Global Compact, θα σας το εξηγήσω, είναι μια πρωτοβουλία που έχει πια κλείσει 15 χρόνια. Είναι η μεγαλύτερη εταιρική πρωτοβουλία με πάνω από 8.000 εταιρείε. Κυρίως ε, προσανατολίζομαστε προς, προς τους επιχειρηματίες και προσπαθούμε να πείσουμε να εργάζονται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και να εμπνεύσουμε, να δώσουμε κίνητρα για να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στη παγκόσμια ανάπτυξη με την ε, ορθή χρήση πόρων και ούτω καθεξής με στόχο πάντα την ανάπτυξη. Αυτή είναι η δική μας θέση. Έχουμε αναπτύξει ένα ρόλο για υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα με υποδείξεις για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα μέσα αυτές οι επιχειρήσεις. Επικεντρωνόμαστε στο ρόλο των επιχειρήσεων μέσα από το διάλογο αλλά και με την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών με 3.000 μη κυβερνητικούς οργανώσεις που συμμετέχουν. Στην προσεχή διαφάνεια και πολύ σύντομα πάλι εισαγωγικά μπορείτε να δείτε ότι η Global Compact και ο ρόλος μας στο θεματολόγιο 2015 στηρίζεται στην αξιολόγηση του γεγονότος ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αλληλεπίδραση αλλά και μακροπρόθεσμο συμφέρον ε, κοινό μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε ιδιαίτερα να, να υπογραμμίσουμε. Βλέπουμε αλλαγές ε, ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με πολλές επιχειρήσεις. Επιλογές οι οποίες συχνά ταυτίζονται με τις επιλογές και της κοινωνίας των πολιτών. Σε ένα πολύ απλουστευτικό γράφημα που σας δείχνω, νομίζω μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Υπάρχει υποστήριξη βεβαίως και ενδιαφέρον επίσης με τη διαπίστωση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξει και η ενεργό συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι πια φραγμός στην ανάπτυξη σε ορισμένε περιοχές, αλλά μπορούν να ε, διαδραματίσουν και ενεργό ακόμη ρόλο για την ε, επίτευξη μιας λύσης. Γι' αυτό, όπως σας λέω, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που έχω αυτή την ευκαιρία να συνεργάζομαι με επιχειρήσεις και να τις ε, καθοδηγώ στη διαδικασία αυτή που έχουμε καταρχάς ευθυγραμμισμένα μέσα από τις διαβουλεύσεις των ΗΕ Εθνών με εστιασμό στα κύρια θέματα και τη συζήτηση στην ομάδα εργασίας και του στόχους και που ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει η δεύτερη φάση που έχει να κάνει με το μηχανισμό υλοποίηση, αλλά όπως είπα εμείς στεζόμαστε κυρίως στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα. 1500 επιχειρήσεις κυρίως έχουμε προσεγγίσει με ευρύτατες διαβουλεύσεις και συνεργασία σε όλο τον κόσμο ακόμα και με επιχειρήσεις της Αφρικής κάποιες αλλά υπάρχουν. Οι διαβουλεύσει αυτέ λοιπόν τι αποτέλεσμα έχουν φέρει, ποια είναι τα κύρια επιτεύγματα και ποια είναι τα κύρια θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Ξεκινώ με τη συζήτηση που γινόταν νωρίτερα για τους στόχους, γιατί με βάση αυτές τις διαβουλεύσεις ε, κάνουμε πολλή δουλειά με τις επιχειρήσεις για να δούμε τι είδους συστάσεις μπορούν να διατυπώσουν οι ίδιες σε σχέση με τους στόχους εδώ βλέπετε τη δική μας προσφορά και υποβολή προτάσεων στο Γενικό Γραμματέα για το τι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες στην επόμενη διαφάνεια, πώς πρέπει να οργανωθούν κατά τρόπον ώστε να είναι ελκυστικές και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι υποστηρίζονται, όπως βλέπετε εδώ, όλες οι παρατηρήσεις, ε, η οικουμενικότητα που έχει γίνει δεκτή από τις επιχειρήσεις και άλλωστε αντιμετωπίζεται και ως μια ευκαιρία για την συγχώνευση ούτως είπε η κοινή αντιμετώπιση θεμάτων που είναι και η καταπολέμηση της φτώχειας και η ανάπτυξη. Ταυτόχρονα θέματα που συζητούνται και στο δημόσιο τομέα, χώρο συζητήσεων αλλά και στις ε, συζητήσεις προχωρούν εκ παραλίλου. Είναι ευκαιρία λοιπόν να συζητηθεί ο ρόλος των επιχειρήσεων στην βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε εδώ μια δομή. Πιστεύω όμως ότι το πιο σημαντικό πρέπει να υπογραμμίσουν ότι υπήρξε συνένεση ότι η καταπόλεμηση της φτώχειας και η ανάπτυξη πρέπει να είναι η πρώτη και κύρια προτεραιότητα και, αυτό, και αυτό το προσπογράφουν και ε, οι επιχειρήσεις καταπολέμηση φτώχειας, λοιπόν, αλλά και η ανάπτυξη πρέπει να γίνει βιώσιμη. Και εδώ έχουμε τις, ε, τα υπόλοιπα βήματα. Ιδιαίτερα λοιπόν προσπαθούμε να οικοδομήσουμε το ρόλο μιας ε, ανάπτυξης όχι ως αυτό σκοπό αλλά ως μέσον βελτίωσης ε, της, των ίσων ευκαιριών, των, της ισότιμης κατανομής του πλούτου και της ανάπτυξης και εδώ τους λοιπούς στόχους που θα είναι και η ειρήνη και η χρηστή διακυβέρνηση που θα αποτελούν ταυτόχρονα και μέσα. Στη συνέχεια έχω καταγράψει, δεν θα μπορείτε να το διαβάσετε ασφαλώς, αλλά γνωρίζετε τους 17 στόχους που έχει προτείνει η Ενικτή Ομάδα Εργασίας Open Working Group, με την οποία συνεργαζόμαστε στενά, που είναι ευπρόσδεκτοι στόχοι και οι οποίοι πιστεύουμε καλύπτουν ευρύτατα τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, από πλευρά των επιχειρήσεων διαπιστώνουμε και εμείς ότι οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για, την, για τις επιλογές των επιχειρήσεων, γιατί και έμπνευση θα προσφέρουν και στόχευση και φιλοδοξίες για το τι μπορούν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις και μπορούν να αποτελέσουν βάση για εταιρικέ σχέσεις διαφορου τομεί σε μια κοινή θεμελίωση χωρίς να χρειάζεται νέα συζήτηση για εταιρικέ σχέσεις και αναζήτηση στόχων και προτεραιοτήτων. Άρα μπορούν να αποτελέσουν αυτοί οι στόχοι με πολύ σημαντική βάση αρκεί να διατυπωθούν κατά τρόπο σωστό και ξέρουμε ότι και οι κυβερνήσεις στην επόμενη χρονιά θα εστιαστούν σε αυτήν την προσπάθεια. Κοιτάμε λοιπόν πώς καλύπτουν συνολικά και οικουμενικά το θεματολόγιο. Έχουμε κάποιες δικές μας θέσεις και ελπίδες για το πώς μπορούν να προχωρήσουν στις παγίωση το επόμενο έτος. Έχουμε τρεις παρατηρήσεις που έχουμε κοινοποιήσει ευρέως. Η μία έχει να κάνει με την ανάγκη για ενοποίηση στόχων. Σε αυτό έχουμε συγκεκριμένε προτάσεις. Μπορούν παραδείγματι να συζητηθούν κάποιοι παράλληλοι στόχοι για την ανάπτυξη, την εκβιομηχάνηση, αλλά που βέβαια συνδέονται και με την ε, καταπολέμηση φτώχειας και την ισόνομη κατανομή του πλούτου. υπάρχει ένας άλλος στόχος που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει ιδιαίτερα με το ρόλο των επιχειρήσεων, χωριστό στόχος ε, για την ε, βιώσιμη κατανάλωση που αποτελεί πολύ σημαντικό μερίδιο νομίζω του θεματολογίου και που καλύτερα θα ήταν να ενταχθεί στην υλοποίηση, κομμάτι της υλοποίηση του 17 λοιπόν μπορεί να ενσωματωθεί και να καταγράφει έτσι το ρόλο μιας βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης ε, ταυτόχρονα βέβαια και ε, χρηματοπιστωτικής διαχείρισης. Έχουμε επίσης ε, το θέμα της αντιμετώπισης της διαφοράς, της χρηστής διαχείρισης, διακυβέρνησης κτλ. Ο ρόλος των επιχειρήσεων τώρα προς την υλοποίηση των ε, βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ένα περίπλοκο γράφημα το οποίο όμως φαντάζομαι θα μπορούσε να εμπλουτίσει τις συζητήσεις σας. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα ε, πέρυσι στην Παγκόσμια Διάσκεψη Γετών. Ε, μάλλον στη διάσκεψη παγκοσμίω ηγετικών επιχειρήσεων για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι επιχειρήσεις ε, και βλέπετε σύντομα κάποιες υποδείξεις για τις προτεραιότητες που εντοπίζουμε εμείς και την ε, συμβολή που μπορεί να προσφέρει το θεματολόγιο 2015 και μετέπειτα. Και εδώ ιδιαίτερα επι επιλέγουμε τις κύριες προτεραιότητες, θέλουμε πιο ευθυγραμμισμένες ε, ε, επιλογές και κίνητρα. που θα ενισχύσουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων στην ε, υποστήριξη της, της βιώσιμης ανάπτυξης και αποφύγει με τον και ζητούμε η επιλογή αυτή να αποτελέσει και σημείο καμπής για τον τρόπο με τον οποίο ε, οι κυβερνήσεις οι ίδιες και οι κρατικές αρχές είτε πρόκειται ε, για τις σχέσεις τους με κρατικές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για τις προμήθειές τους ή τους διαγωνισμούς ή την κατανάλωσή τους, να έχουν και αυτές αντίστοιχη προσέγγιση. Καλούμε δηλαδή και τις, επιχει... και τις ε, κυβερνήσεις, τα κράτη, να αναπτύξουν ρόλο ηγετικό στο βαθμό που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στις επιλογές αυτές και έτσι μπορούν να ακολουθήσουν και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν περισσότερε εταιρικέ σχέσεις των εμπλεκομένων φορέων. Οι εταιρικέ σχέσεις ιδιαίτερη σημασία έχουν για τα Ηνωμένα Έθνη όταν ε, βλέπουμε ότι είναι περισσότερες ε, οι ανάγκες για εταιρικέ σχέσεις ε, σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που επί παραδείγματι μπορεί να μην έχουν αρκετούς πόρους, γραμματιακή υποστήριξη και ούτω καθεξής. Εκεί μπορούμε να, να εντοπίσουμε τις ανάγκες για εταιρική σχέση αλλά και στο συντονισμό των προσπαθειών στο με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτές είναι οι εταιρικέ σχέσεις και βέβαια εδώ το θέμα της λογοδοσίας από τις εταιρικέ σχέσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία στο θεματολόγιο για την ανάπτυξη μετά το 2015. Μπορούμε να διατυπώσουμε κάποια μέτρα ε, οι προδιαγραφές για διαφάνεια στις σχέσεις και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής με ένα εθελοντικό, με ένα εκούσιο σύστημα αξιολόγησης της διαφάνειας. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ, διαφάνεια, λογοδοσία στον ιδιωτικό τομέα, στην εμπλοκή και δέσμευση του ιδιωτικού τομέα και εδώ θέλουμε να πούμε ότι η συζήτηση δεν χρειάζεται να ξεκινήσει εκ του μηδενός. Έχουμε ήδη αλλάξει σε πολλά πράγματα. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία 10-15 χρόνια και θα πρέπει να αξιοποιηθούν και η διαφάνεια η εταιρική και η λογοδοσία και τα συστήματα πιστοποίησης. Υπάρχουν ήδη. Όλα αυτά είναι μέσα, αυτό έχουμε να πούμε εμείς, μέσα τα οποία ε, επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να καταστούν πολύ πιο θετική δύναμη για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αντί λοιπόν για νέα μέσα πρέπει να χτίσουμε πάνω στις υφιστάμενες ιδέες που υπάρχουν. Κάποια κενά έχω εντοπίσει ως προς την διαφάνεια για τις εταιρικέ σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα και κάτι άλλο στο οποίο συνεργαζόμαστε με το Παγκόσμιο Επιχειρησιακό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αξιολόγηση αντικτύπου έτσι ώστε να καταγράφεται η πρόοδο σε σχέση με τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, να καταγράφεται ποιο τούβλο στο οικοδόμημα έχει επιτευχθεί και ενδεχομένως σε ποιο σημείο υπήρξε πρόβλημα από πλευράς των δράσεων των επιχειρήσεων πάντα σε, με μέτρο τους αναπτυξιακούς στόχους ε, ώστε να δούμε που υπάρχουν ελλείψεις και, και να ε, ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου αλλά θα ήθελα κλείνοντας να πω μερικά λόγια για τη χρηματοδότηση, για τον οικονομικό σκέλος. Πριν από κανένα δύο μήνες μαζί με άλλους ε, θεσμούς, φορείς ε, του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για την ε, ιδιωτική βιώσιμη χρηματοδότηση, όπου όλοι να γνωρίζουν τον κέριο ρόλο της διαχείρισης των κονδύλιων και αυτό το λέμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει όχι να υποκαταστήσουν αλλά να συμπληρώσουν τα εφιστάμενα μέτρα. 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια πρόσθετων επιχειρήσεων λένε ορισμένοι ότι χρειάζονται ε, και ότι μπορούν να, να συμπληρώσουν τους υφιστάμενους πόρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να, νέα, να αναστήσουμε νέα ποσά, νέα επενδυτικά μέσα, αλλά αντιθέτως σημαίνει ότι υπάρχουν υφιστάμενες ροές επενδυτικές, τις οποίες απλώς θα πρέπει να ε, αντλήσουμε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως να αλλάξουμε και τη ροή τους. Αυτά και θα είχα κάποιες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, αλλά επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε τον ε, ιδιωτικό τομέα λεπτομερώες περιττέρω. Οπότε δεν έχουμε χρόνο. Ας ε, επικεντρωθούμε στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης προς το παρόν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των ερωτήσεων. Μέχρι στιγμής μόνο ένα άτομο έχει ζητήσει τον λόγο, αλλά να, τώρα είναι περισσότεροι. Ο πρώτος ομιλητής, ο κ. Νόιζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στα προβλήματα που διαπιστώνω σχέση με τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Ήταν ε, μια υπόθεση επιτυχίας η αναπτυξιακή στόχη αυτή, γιατί ήταν πολύ σαφής η διατύπωσή τους και ε, μπόρεσαν να είναι κατανοητοί για τους θωρινούς στόχους, ε, τους 17 αυτούς στόχους που είναι ασαφείς, που είναι δύσκολο να δει κανείς στο σύνολό τους, θα πρέπει πιστεύω να κάνουμε μια προσπάθεια, να τους ε, συνοψίσουμε και να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ στόχευσης, μεταξύ προβλεπόμενων στόχων και μεταξύ υλοποιούμενων στόχων. Και επίσης Κύριε Πρόεδρε, στα όσα είπατε για την προσέγγιση στα ανθρώπινα δικαιώματα, θέλω και εγώ να υπογραμμίσω ιδιαίτερω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η πιο ισχυρή εμπλοκή και επέμβαση στο θέμα των δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ακόμα σαφέ το πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σε πολιτικό επίπεδο, σε ύψιστο επίπεδο, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσει, μπορούμε νομίζω να διατυπώσουμε σαφεί θέσει προ τον Κιμούν και να στηρίξουμε τις προσπάθειές του. Αυτή λοιπόν τη διάσταση των δικαιωμάτων θέλουμε να υποστηρίξουμε και ιδιαίτερα να διατυπώνονται οι στόχοι έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της υλοποίησης του σε κάθε κράτος. Η κυρία Σλάιν. ο ορισμός ε, του χρονοδιαγράμματος μετά το 2015 είναι σημαντικός γιατί βρισκόμαστε σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτόν στο οποίο έγιναν αντικείμενο διαπραγμάτευση οι στόχοι τη ηλιτία. Είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο για να λάβουν τι νέε αυτέ προκλήσει. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καθοριστικό ρόλο, θα πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια να μιλήσει με μία και μόνο φωνή για να μπορέσει να συμβάλλει καλύτερα σε αυτή τη συζήτηση. Από αυτή την άποψη, οι προσδοκίε προς τη νέα Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο είναι πάρα πολλέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Τζέφερσον, γιατί πιστεύω ότι έθιξε τρία σημαντικά σημεία. Το θέμα της παγκοσμιότητας αυτών των κοινών ευθυνών αλλά και το θέμα των ανισοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο νέο πλαίσιο να υπάρχει υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχο που αφορά την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Γιατί πιστεύω ότι με αυτή την πρόκληση έχουν σχέση πολλά θέματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Όπως οι συγκρούσεις που ανοίγονται, το πρόβλημα τη της ενέργειας, αλλά και το πρόβλημα της μετανάστευση. Θα ήθελα να καταλάβω αν θα είναι δυνατόν να διατηρήσουμε στο κέντρο της σκέψης μας στόχους που αφορούν τα αναπαγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα στην υγεία. Αν θα είναι δυνατόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Πιστεύω ότι η στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι λιγότερο νεφελώδης και θα πρέπει να γίνει και μία αναφορά στο θέμα της ε, φτώχειας και της ε, περιγενετικής υγείας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Γκέρενς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω για τους δείκτες. Στο τέλος της διαδικασίας θα έχουμε δείκτες που θα μας πούν για την ποιότητα, την καθαρότητα, την ποιότητα, την υγεία, την διακυβέρνηση κλπ τότε θα έχουμε μια συνολική άποψη για έναν κλάδο, μια, ένα τομέα, μια χώρα, μια περιφέρεια. Μπορούμε να πούμε λοιπόν τότε αν, αν ε, υπάρχει υπαρκής πρόοδο, αν αυτά είναι ικανοποιητικά. Για, το, για τη δική μας, για μας Ποιοι είναι οι δείκτε που θα κινητοποιήσουμε για να μετρήσουμε την προσπάθεια που καταβάλουμε. Είμαστε κομμάτι της λύσης ή, της, ε, ή του προβλήματος. Επιμένω, διότι υπάρχει μια παράλογη κατάσταση όπου οι δείκτες που ζητώνται για τους δείκτες της βιώσιμης ανάπτυξης ε, ο καθένας έχει την τάση να χρησιμοποιεί τους δείκτες που τον <laughs> βολεύουν και που μπορεί να τους ε, πετύχει με ελάχιστη προσπάθεια. Και άρα δεσμευόμαστε να επιβάλλουμε κριτήρια που θα είναι τα ίδια για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδάλλως, η σύγκριση των εθνικών προγραμμάτων δράσης για την πρόθεση των στόχων που θα προκύψουν από αυτή την προσπάθεια δεν θα έχουν κανένα νόημα. Καλή είναι η παρακολούθηση, και η, αλλά η συνεκτικότητα της πολιτικής και ο συντονισμός είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να τα ε, θέσουμε από τώρα. Ευχαριστώ κύριε Βάνη. Κυρία Πρόεδρε, τέσσερα σημεία, τέσσερις ερωτήσεις. Καταρχάς η αρχή της παγκοσμιότητας. Βεβαίως θα πρέπει να προωθήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για περιορισμό της ένδυας σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Δεύτερον, περιορισμοί των πόρων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το παγκόσμιο ΑΕΠ μετά από 50 χρόνια θα είναι 5 φορές υψηλότερο από ό,τι τώρα και στις χώρες του ΩΣΑ 3 φορές υψηλότερο. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό να υπάρχει αυτό, να συμβεί κάτι τέτοιο τα επόμενα χρόνια. Ακόμα και όταν οι τεχνολογίες βελτιώνονται, υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν τους σπόρους και το περιβάλλον. Τρίτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καλή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, όταν η βασική μας στόχη είναι η μείωση της στόχιας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ένας από τους τρεις επιλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η κοινωνική βιωσιμότητα. Και η βάση για την κοινωνική βιωσιμότητα είναι το ε, σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την καλή διακυβέρνηση. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για κάθε είδους ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν μία βάση για να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες με βάση τις αρχές για το 90, ε, ε, ε, τις που έχουμε θέσει. Το πρόβλημα είναι ότι έξι, έχουμε έξι συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τη μείωση της ένδυας. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου αντλούσαμε συνέχεια δημόσιο χρήμα σε μια προσπάθεια να επηρεάσουμε αυτούς τους στόχους. Βεβαίως όλα αυτά ήταν θετικά, αλλά η πιο αποτελεσματική μείωση της φτώχειας επετέφθη σε χώρες με ε, γενική ε, ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Κάναμε μία προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η οικονομική ανάπτυξη. Χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα... Ε, ε όλη η χρηματοδότηση. Όταν συζητάμε λοιπόν τους νέους στόχους δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον στόχο υπαριθμών 1 που είναι η εκρίζωση της ακραίας φτώχειας και της πείνας. Αλλά παράλληλα παραμελήσαμε την ανάπτυξη της γεωργίας για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για τους στόχους και τα μέσα και το πόσα θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους βασικούς στόχους της μείωσης της ε, ε, φτώχειας και της ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Η στόχη τη Αφρικανική Ένωση είναι πάρα πολύ καλή κατά την άποψή μου. Είναι απτή, είναι συγκεκριμένη. Και υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα που προβλέπετε. Θα θέλαμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια για αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Α, μία ερώτηση, αλλά πάρα πάρα πολύ σύντομη, γιατί έχουμε μόνο 10 λεπτά, 7 λεπτά και θέλουμε να τελειώσουμε στην ώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να επιμείνω όσο προς την ε, κατάσταση που παρατηρείται κάθε μήνα, κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο που διαπιστώνουμε ότι το οικονομικό, κοινωνικό ε, και ε, περιβάλλον και τα θέματα ασφαλείας αλλάζουν ε, με τρόπο εντυπωσιακό. Τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε αντιμέτωποι με διαφορετικές αλλαγές αυτού του περιβάλλοντος και αυτό έθεσε πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόοδό μας. Θα ήθελα να επιμείνω για ως προς το απόθεμα που θα πρέπει να δημιουργηθεί για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο προγραμματισμός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα πράγματα δεν είναι όπως είχαν. Θα πρέπει να προγραμματίζουμε εκ των προτέρων και να προλαμβάνουμε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, γιατί ζούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον το οποίο αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πράτα, θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Παρακαλούμε θερμά τους διερμηνείς να παραμείνουν για 5 ή 6 λεπτά πέραν του ωραρίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλια από τους συναδέλφους από την οργάνωση Concord. Καταρχάς ήθελα να διαβεβαιώσω και εσάς και την Επιτροπή ότι η θαυμάσια συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα με την κοινωνία των πολιτών μέσω της Ευρωπαϊκής ε, task force ε, θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί και η θαυμάσια συνεργασία με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Παριβάλλοντος. Βεβαίως ε, πρόκειται να οριστεί το νέο κολέγιο επιτρόπων, αλλά είμαι αισιόδοξο ότι θα συνεχιστεί το έργο των προηγούμενων επιτρόπων. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην Επιτροπή. Η συνεργασία αυτή συμπεριλαμβάνει και τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Εξωτερικής Δράσης από τη μία πλευρά, αλλά και το Συμβούλιο. Τα θέματα αυτά πάντοτε συζητήθηκαν στο Συμβούλιο στην συνάντηση τζάμπο των τριών επιτροπών ε, που συναντώνται πάντα ε, μαζί ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ανάπτυξης ε, περιβάλλοντος. Τώρα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε επικεφαλής αυτής της συζήτηση και θα συνεχίσει να το κάνει στα πλαίσια και μετά το 2015 γιατί συμφωνούμε ότι είναι καθοριστική σημασία κάτι τέτοιο. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης ε, του χρόνου είναι σαφές ότι η συνάντηση μετά το 2015 ε, θα είναι εντελώς ε, διαφορετική και δίχως άλλο μας βρίσκει σύμφωνο η συμμετοχή σε όλες αυτές τις διοργανώσεις του Κοινοβουλίου καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Οι ομιλητές μας παρακαλώ. Ο κύριο Τζέφερσον. Πολύ τρία λεπτά. Θα είμαι γρήγορο. Χωρί να επιδιώξω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα, δύο-τρει σκέψει. Πρώτον, βασική σημασία, η μετρήσιμότητα. Και αυτό απαντά ίσω και στι δύο ερωτήσει. Δύο είναι τα ζητήματα. Πρώτον είναι η παρουσίαση των στόχων με τους οποίους καταλήγουμε όταν τελειώσει η τεχνική δουλειά θα πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό, ώστε ο κόσμος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Και επίσης, επανερχόμενος σε αυτό που ονομάζουμε στη γλώσσα μας η προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει συμμετοχή δηλαδή. Αυτοί τους οποίους επηρεάζει η πολιτική οφείλουν να συμμετέχουν στο, εάν και, στο τον έλεγχο του εάν και κατά πόσον οι πολιτικές αυτές κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Και στο χώρο μας υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν δουλέψει με τη συμμετοχή των πολιτών για την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των δημοσίων ε, υπηρεσιών μέσω smartphones και το θέμα των εμποδίων στην ε, διαφθορά κλπ. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε για την μετρησιμότητα των, ε, ε της των στόχων της χιλιετίας και αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αυτούς που συμμετέχουν. Τώρα, το θέμα της ανισότητας. Σπανίως στο παρελθόν έχει υπάρξει τέτοια συνένεση ε, σε όλο το πολιτικό φάσμα για το θέμα αυτό της ανισότητας το οποίο πραγματικά έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και αυτό επηρεάζει τους πάντες δηλαδή κινδυνεύει ο κοινωνικός ιστός, ο οικονομικός ιστός και όταν το Δούνου του και οι τα πολιτικά κόμματα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις συμφωνούν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει για την αντιμετώπιση της ανισότητας. Όλοι ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα, τι θα κάνουμε περί αυτού και επ' αυτού πρέπει να δουλέψουμε. Φορολογικά συστήματα, παράνομες ροές, ε, ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κλπ. Ευχαριστώ. Ε, εν συντομία επίσης για κάποια παρόμοια θέματα. Η ισότητα. Στο τέλος της ε, περσινής διαδικασίας θεωρήσαμε ότι ζητήσαμε από τις επιχειρήσεις ε, να υποστηρίξουν αυτούς τους, τους στόχους της μείωσης της ένδυας και της ισότητας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει γενική εκτίμηση ότι όχι μόνο η περιόριση της ε, ε, ένδυας αλλά και τα θέματα της συμμετοχή συμμετοχής είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεύτερον, όλοι συμφωνούμε και εμείς υποστηρίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα πρέπει να δουλέψουμε από αυτό που κάνουμε τώρα σε κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο και μετρήσιμο η αρχιτεκτονική που έχουμε κατά νου και εμείς και άλλοι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τους ίδιους τους στόχους. Δηλαδή να, να εμπνέουν και να είναι εύληπτοι. Όσον αφορά τώρα τα αντικειμενικά αποτελέσματα πρέπει κανείς να είναι, να, πρέπει να είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα. Ιδάλλως δεν, θα δεν έχει νόημα να ε, εμπνέουν οι στόχοι. Ε, υπάρχει ένα θέμα με τους ε, δείκτες, υπάρχει η Στατιστική Επιτροπή του ε, ΟΗΕ, υπάρχει ε, το δίκτυο των βιώσιμων λύσεων που επικεφαλής είναι η ΣΑΚΣ κτλ. Αλλά το θέμα ε, των αναπτυξιακών στόχων είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές ομάδες και διαφορετικοί εμπλεκόμενοι και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και με τις επιχειρήσεις και με τους επενδυτές. Δηλαδή έχουμε κοινωνικούς στόχους, δείκτες και Ποιο είναι ένας ε, ουσιαστικό τρόπος που να εξυπηρετεί και τι επιχειρήσει να μετρηθούν όλα αυτά. πώ πώς μπορεί να μετρηθεί, τι έχει, πώς επηρεάζει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που θέλουμε να ενθαρρύνουμε και να το υποστηρίξουμε ώστε να αναπτυχθεί. Πέραν αυτού, είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτο ότι θα κάνετε εσείς συζήτηση για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Εμείς θεωρούμε ότι ε, ο ρόλος του θεματολογίου ανάπτυξης μετά το 2015 είναι σημαντικός και το θέμα είναι αν είμαστε όχι υπέρ κατά της εμπλοκής των επιχειρήσεων, αλλά δούμε με πρακτικό τρόπο πώς θα μειώσουμε την αρνητική επίπτωση που έχουν κάποιες επιχειρήσεις και πόσο όλα αυτά θα γίνουν μια θετικότερη δύναμη για την ανάπτυξη. Να αποφύγουμε τη συζήτηση που εξακολουθεί σε μερικούς χώρους μερικές φορές υπέρ κατά όλοι. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι πόροι, είναι τεράστια η επίπτωση. Πρέπει λοιπόν να ε, επισπεύσουμε μέσω αυτού του θεματολογίου την μετάβαση προς τα εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που μας θύμισαν, γιατί πολύ συχνά συνηθίζουμε να μιλάμε για τον αναπτυσσόμενο κόσμο και τον αναπτυγμένο κόσμο, όπως είπατε όλοι. Ε, ένας είναι ο κόσμος και όλοι τον μοιραζόμαστε και πρέπει να το κάνουμε σωστά, ιδάλλως τα προβλήματα θα, θα διαπεράσουν τα πάντα, όλα τα μέρη του κόσμου. Και έτσι αυτό ίσω να είναι η ουσιαστική διαφορά από τι προηγούμενε συζητήσει για την ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπω σα είπα και πριν, ξεκινάμε μόλι τώρα τη συζήτηση. Θα έχουμε μια έκθεση ιδία πρωτοβουλία. Όλε οι πολιτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου θα συμμετέχουν. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μα του επόμενου μήνε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ του ομιλητέ. Uh, και ε, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρωινή συζήτηση. Θα επιστρέψουμε στις 3 για τη συζήτηση για τον προπολογισμό και κατόπιν θα έρθει η Επίτροπος Γεωργίευα να μας μιλήσει για την ανθρωπιστική βοήθεια και τα πολύ σοβαρά θέματα που είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Everything is here. Yeah, we stay here, of course. Yeah, we, stay here. Normally committees take place in Πάλι εδώ θα είμαστε στην ίδια αίθουσα. Ευχαριστώ και του διερμηνείς.